Ο πρόεδρος. Αρχίζουμε λέει. Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy megnyissam a délutáni találkozást. Σας καλωσορίζω στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω ουγγρικά. Προτού όμως ε, κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας για την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές του Bundestag, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια κυρία από τη Σλοβακία, την κυρία Πατσάνοβα, η οποία έχει υποβάλει μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά που συνδέεται με τον δολυφέντα δημοσιογράφο. Να πω και κάτι στα σλοβακικά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να την ακούσουμε. Να καλωσορίσω τώρα τους ε, εκπροσώπους του Bundestag. Έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Βέρντ ε, εκ μέρους του Τσεντεού, τον κύριο Σβάρτσε, τον κύριο Μούλερ, τον κύριο Βίλε, τον κύριο Ούλριχ και τον κύριο Έμπινγκ, τον κύριο Χούμπερτ και εκ μέρους της αριστεράς του Κόμματο Αριστερά έχουμε μαζί μα τον κύριο Ζόρεν Πέλμαν. Ελπίζω να τα προέφερα σωστά τα ονόματα, αν όχι να με συγχωρήσετε. Σα καλωσορίζω θερμότατα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι μία από τις σημαντικότερες ε, υποχρεώσεις μας να φροντίζουμε την άμεσή μας επαφή με τους πολίτες από τα 28, 28 κράτη-μέλη ε, γνωρίζετε ότι κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται σε εμάς σε περίπτωση που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Η Επιτροπή μας κάθε μήνα συνεδριάζει μία φορά και ξέρετε ότι σε κάθε συνεδρίαση ε, επεξεργαζόμαστε μια πλειάδα αναφορών. Σήμερα στη σημερινή μας συνεδρίαση είχαμε πολλές γερμανικές αναφορές. Τέσσερις από αυτές εντάσσονταν ε, στην ε, θεματική κατηγορία του περιβάλλοντος. Μάλιστα είχαμε και μια ψηφοφορία σήμερα το πρωί που αφορούσε τη Γερμανία. Έχουμε λοιπόν μια ειδική ημέρα αφιερωμένη στη Γερμανία, αν θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βέλε για λίγα λεπτά. Και σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι από τον Bundestag, βουλευτές της Γερμανίας, να μου κάνετε ένα νόημα, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζακ, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι της Ευρώπης. Εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών της Γερμανικής Βουλής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θερμά σας λόγια, για το καλωσόρισμα αυτό και για την δυνατότητα που μας δίνετε να συμμετέχουμε εδώ στη συνεδρίασή σας σήμερα. Τελευταία ε, επίσκεψη ε, της Επιτροπής Αναφορών από τη Γερμανία έγινε το 2015 υπό την αιγίδα με επικεφαλή στην κυρία Στάινκε. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε σήμερα αυτό το διάλογο μαζί σας διότι ε, μας ενδιαφέρει η εντατικοποίηση ε, των σχέσεων ιδίω των Επιτροπών Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Το 2007, για παράδειγμα, υπήρχαν 20 αναφορές που διαβίβασε το, το Γερμανικό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρσι ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 120. 120 δηλαδή αναφορές διαβιβάσαμε ως Γερμανικό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από αυτό και μόνο φαίνεται ότι οι ναι. σχέσεις μας είναι όλο και πιο στενές και ότι Εργαζόμαστε ακούραστα όλοι μας για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει την ε, αρμοδιότητα, τα κρατήδια, τα κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος όλων μας στη δουλειά μας είναι να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών. Γιατί νομίζω ότι στους πολίτες, άλλωστε τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποιος και με ποιον τρόπο θα διευθετήσει τα θέματα του, θέλει να διευθετηθούν για να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο κράτος και στη διοίκηση. Μια ιδιαίτερη αναφορά βεβαίως αφορά την αλλαγή της ώρας. Αν και δεν, ίσως δεν είναι το σημαντικότερο θέμα, αλλά ε, είναι ένα θέμα το οποίο κινητοποιεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάνω από 500 ε, άνθρωποι συμμετείχαν στην έρευνα την ε, διαδικτυακή που ε, διοργανώσαμε εμείς. Νομίζω ότι και εμείς αύριο στην Επιτροπή Αναφορών του Γερμανικού Κοινοβουλίου έχουμε μια τέτοια αναφορά την οποία θα συζητήσουμε. Οπότε θα ήταν πραγματικά ε, πολύ χρήσιμο αυτή τη στιγμή να βρεθεί μια έξυπνη λύση στο πρόβλημα αυτό και όχι να επιστρέψουμε φυσικά στην εθνική ρύθμιση του θέματος αυτού, της θερινής ώρας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ για το κοινό μας έργο όσον αφορά τις αναφορές που σχετίζονται με την Ευρώπη και ιδίως τη Γερμανία αφού είμαστε εκπρόσωποι του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν και ε, θα βεβαίως ε, σας κάνουμε κάποιο νόημα αν θέλουμε να ξαναπάρουμε το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους του Γερμανικού Κοινοβουλίου αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρόεδρος τα είπε όλα. Όχι. Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον Γερμανό συνάδελφό μας εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γερμανική υπόθεση η σημερινή μας συνεδρίαση. Φαίνεται και από τους συμμετέχοντες. Και βλέπετε, κατευθείαν δόθηκε ο γερμανικός τόνος. Πάμε στη δουλειά. Στην ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να πω και εγώ ότι είναι πολύ θετικό και χρήσιμο το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ. Είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιτροπών ε, αναφορών. Εμείς λοιπόν είμαστε οι πλησιέστεροι στους πολίτες επιτροπή. Είμαστε κάποιες φορές η έσχατη λύση, είμαστε οι καλοί αν θέλετε ε, γιατί επεξεργαζόμαστε πραγματικά θέματα που απασχολούν πάρα πολύ τους ε, πολίτες μας στρέφονται προς εμάς πολύ συχνά οι πολίτες μας για να λυθούν τα προβλήματά τους το ίδιο βεβαίω ισχύει και για το, για το Γερμανικό Κοινοβούλιο και την αντίστοιχη Επιτροπή Αναφορών μια διαφορά μας με την Επιτροπή Αναφορών είναι το γεγονός ότι επεξεργαζόμαστε απευθείας τις αναφορές μπορεί μάλιστα ο κάθε πολίτης να προσέρχεται εδώ προσώπο στην Επιτροπή για να παρουσιάσει την υπόθεσή του. Καλό είναι αυτό, χρονοβόρο βέβαια και από την άλλη μεριά, αλλά ε, ίσως είναι και αυτό μια ιδέα που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από το Βερολίνο. Τρίτο, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, καλύτερα πλέον. Το είπε και ο Πρόεδρος. Ε, πολύ συχνά λαμβάνουμε αναφορές ή διαβιβάζουμε εμείς ε, ε, αναφορές σε εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, δηλαδή να καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος έχει την εμπνοδιότητα, αναλόγως του θέματος κάθε αναφοράς, προκειμένου να μπορούν να επεξεργάζονται και να βγαίνουν και συμπεράσματα ε, αλλαγή θερινής ώρα και κατάργηση θερινής ώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αποδεικνύει ότι οι Βρυξέλλε δεν ασχολούνται μόνο με τα πολύ μεγάλα θέματα αλλά και με τα καθημερινά των πολιτών. Και εδώ είναι ένα θέμα στο οποίο πραγματικά ε, στάθηκε επικεφαλής η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς το ανακοινήσαμε αυτό το θέμα εξ αρχής πολλές φορές. Έφτασε τελικά μέχρι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και επέβαλε πρόταση. Και είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να βοηθούμε και να βελτιώνουμε ακόμα και τις καθημερινές πλευρές ε, της ζωής των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ας περάσουμε λοιπόν στα συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε πέντε αναφορές, έχουμε ένα πακέτο. Πρώτο, ο Βάλτα Μπέχτα, αναφορά 0533-2014, 1735-2013 μάλλον για την μόλυνση δύο ποταμών αναφορά 0533 του 2014 για, την, ε, για το λατούχο νερό στο Ομόσπονδο τη της ΣΕΣΙΣ. Μια τρίτη αναφορά έχει να κάνει με τα λατούχα διαλύματα από τη βιομηχανία στον ποταμό Μπαβέζα στη Γερμανία. που επιβαρύνει το περιβάλλον και τέλος ε, μία ε, αναφορά από τον Πέτα Ζιλμπανάγκελ 1287 για τη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στη Γερμανία. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παρόντες ή αναφέροντες, αλλά επειδή έχουμε web streaming, θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της DJ Envy, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, να εκφράσουν την άποψή τους για, τις, ε, για την κάθε μία από τις ε, αναφορές αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά την τελευταία επικαιροποίηση, πριν από ένα χρόνο της Επιτροπής, οι επιπαραβάσεις διαδικασίες που έχουμε με, σε με αυτές ε, τις αναφορές είναι ακόμα ανοιχτέ. Υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται ήδη στη Γερμανία. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τώρα έχουμε λάβει όλη την τεκμηρίωση και τα δεδομένα από την ε, ενδιαφέρουσα χώρα, τη Γερμανία και η εξολόγηση της Επιτροπής Και το δεύτερο πρόγραμμα διαχείρισης της λικάνης απορροής ε, των ποταμών έχει προχωρήσει κατά πολύ. Τελειώνουμε το τεχνικό μας έργο ε, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμμετοχή μεταξύ των 28 κρατών μελών, γιατί έχουμε κάνει ισότιμη διάγνωση για όλα τα κράτη-μέλη. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, αυτό το έχουμε ολοκληρώσει μέσα στον επόμενο μήνα, θα μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το δεύτερο πρόγραμμα διαχείριση ε, των νεκρών απορροή ποταμού και για αυτέ τι περιπτώσει. Και σε εκείνη τη χρονική στιγμή θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε και την Επιτροπή σα. Ευχαριστώ. Άρα βρίσκεται ε, σε εξέλιξη η διαδικασία. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους από τον Bundestag αν θέλουν να τοποθετηθούν. Το μικρόφωνο του ομιλητή δεν είναι αναμένο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς ε, να σας πω ότι είναι τιμή μου το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ ε, για ένα θέμα που αφορά και την εκλογική μου περιφέρεια και εγώ ε, κατάγομαι από την ΕΣΥ. Το πρόβλημα είναι μπροστά στην πόρτα μου δηλαδή. Έχω όμως και μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την K+S, ε, με πάρα, πολύ, πάρα πολλές θέσεις εργασίας που προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της απασχόλησης. Αυτό είναι πάντοτε πολύ μεγάλη πρόκληση. Για μένα είναι σαφές πάντως ότι το, η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα είναι η βάση, η, καθορίζονται εκεί οι βασικές διατάξεις που θα πρέπει να τηρούνται. Από αυτή την άποψη ε, ασχολούμαστε και ε, βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με την επιχείρηση. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και η ίδια η επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο να λύσει το πρόβλημα που υπάρχει. Λύση η οποία θα καταλήξει στο ότι η επιβάρυνση του, του ποταμού Βέρα και του πεταμού Βίζε θα μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να, τηρεί, να τηρείται πλέον η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ασκήσει πίεση στην ε, εταιρεία αυτή και από αυτή την άποψη η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θετικό προκειμένου να ασκηθεί πίεση και να βρεθεί λύση. Ε, λύση η οποία όπως είπα θα ε, επιτυχάνει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Ε, προφανώς ε, καλά τα είπε ο συνάδελφο από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ε, ευρωπαϊκοί νόμοι που πρέπει να εφαρμόζονται. Τώρα αν γίνεται αυτό καλά ή λιγότερο καλά, αυτό ε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Κάποιες φορές δεν εφαρμόζεται σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, λάβαμε κάποια, ε, ε, έλαβε μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια καταγγελία, μια αναφορά. Τουλάχιστον όμως έχει ξεκινήσει ένας, ένας διάλογος με την επιχείρηση και από ό,τι ακούμε φαίνεται ότι και η ίδια η εταιρεία έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται. Δράση ανέλαβε και η τοπική αρχή του κρατηδίου ε, βρισκόμαστε από ό,τι φαίνεται προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα να ε, κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή ώστε να λάβουμε και τις τελικές ε, οριστικές πληροφορίες από την Κομισιόν και να μας διαβεβαιώσουν και από την πλευρά της Κομισιόν ότι πραγματικά το θέμα έχει πλέον διευθετηθεί, έχει επιληθεί γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να προστατευτεί το περιβάλλον εκεί της περιοχής. Συζητήσαμε κάτι αντίστοιχο και το πρωί αφορούσε βεβαίως την ε, καθαρότητα του αέρα και τη σχετική οδηγία. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μεταφέρετε το μήνυμα στο Βερολίνο, λοιπόν. Ε, αυτό που θέλω εγώ να στείλω στο, Βερολίνο. Όταν αποφασίζετε και θεσπίζετε ευρωπαϊκή νομοθεσία, και συμμετέχουν οι συνομοθέτε, τα κράτη-μέλη, οι κομισιόν, τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι αυτή η νομοθεσία θα πρέπει στη συνέχεια και να εφαρμόζεται. Διότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο να θεσπίζεται νομοθεσία εδώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμω με πολύ μεγάλη δυσκολία ή και καθόλου δεν εφαρμόζεται μετά στα κράτη-μέλη. Ε, ως προς τις ε, οριακές τιμές που ε, καθορίζονται στην οδηγία πραγματικά είναι πολύ δύσκολες αλλά εγώ το μόνο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω από αυτό είναι ότι θα έπρεπε τότε τα κράτη-μέλη στη διαδικασία θέσπισης του συγκεκριμένου νομοθετήματος να είχαν παρέμβει και να είχαν επιδείξει σοβαρότερη στάση ώστε να μπορεί η νομοθεσία στην οποία θα καταλήγουμε κάθε φορά να εφαρμόζεται και από τους αρμόδιους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πρόεδρος, ε, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Επομένως, σημειώνουμε τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρίσκεστε λοιπόν στο μέσο μιας διαδικασίας, συνεχίζεται ο διάλογος, ελπίζουμε ε, με κατεύθυνση και ορίζοντα την εξέβρεση λύσης. Είμαστε στη διάθεσή σας, θα είμαστε και σε συχνή επαφή. Μόλις ε, ανακύπτουν νέα δεδομένα και αποτελέσματα θα είμαστε ενήμεροι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ε, αναφορά, την 1025, την 0793 του Μανφρετ Χέσνερ και τρίτη αναφορά σε αυτό το μπλοκ αναφορών που θέλουμε να συζητήσουμε είναι η αναφορά 0819 του 2017 ε, του TH Γερμανική ηθαγένεια σχετικά με την ε, μόλυνση νητρικών αλάτων του πόσιμου νερού στη Γερμανία. Δεν είναι μαζί μα δυστυχώ οι αναφέροντες, μας παρακολουθούν όμως από το ίντερνετ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μα παρουσιάσει τη θέση της Γενικής διεύθυνση περιβάλλοντο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα των νητρικών που μολύνουν τα ύδατα. Η υπερβολική ποσότητα βλάπτει το περιβάλλον, έχει επιπτώσει στην υγεία και τέλος η διαδικασία καθαρισμού είναι, κοστίζει πολύ. Από το 1991 υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια οδηγία που έχει στόχο να μειώσει την ε, μόλυνση από τα νητρικά ε, λόγω αγροτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στη Γερμανία και την εφαρμογή της οδηγίας, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Γερμανία υπέβαλε ε, κάποια στοιχεία το 2012. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξε αυξημένη ε, μόλις των υπόγειων υδάτων από νητηρικές ενώσεις και από άζωτο, από άζωτο, και ο στόχος είναι να μειωθεί η μόλυνση των υδάτων από ε, το άζωτο, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη. Η Γερμανία επίσης δεν ε, έλαβε τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα που σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να ληφθούν όταν γίνεται προφανές ότι η ποιότητα του νερού δεν έχει βελτιωθεί. Έτσι λοιπόν το 2016 η Επιτροπή ε, η Ευρωπαϊκή στο δικαστήριο ε, και τα δεδομένα που ε, υποβλήθηκαν για την επόμενη περίοδο 2012 και 2015 έδειξαν ότι δεν υπήρξε επαρκής ε, βελτίωση στον τομέα της μόλις από το άζωτο. Σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018, το δικαστήριο απεφάνθη ότι η Γερμανία δεν είχε συμμορφωθεί με την οδηγία γιατί είχε αποτύχει να ε, λάβει τα πρόσθετα μέτρα. Όταν πλέον ήταν προφανές ότι τα μέτρα στο τρέχον τότε πρόγραμμα ήταν ανεπαρκή. Στο μεταξύ, το 2017 η Γερμανία εισήγαγε τη νέα νομοθεσία για τα λοιπάσματα, η οποία ε, τέθησε εφαρμογή. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η απόφαση του δικαστηρίου του 2018 αφορούσε την προηγούμενη νομοθεσία την νομοθεσία που ήταν ενισχύ μέχρι τη νέα νομοθεσία σχετικά με τα λοιπάσματα, η οποία ε, τέθηκε σε αρμογή το 2017. Άρα λοιπόν τώρα η Επιτροπή αξιολογεί τη νέα νομοθεσία υπό το φως της απόφασης φυσικά του δικαστηρίου ενώ παράλληλα είμαστε σε επαφή με τις Ομοσπονδικές Αρχές της Γερμανίας για να συζητήσουμε πώς ε, προτίθεται να συμμορφωθούν με την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στρέφομαι προς τα μέλη του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την πρόσκληση βεβαίω και για το γεγονό ότι έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ. Εξ όσων γνωρίζω, χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για να εμφανιστεί στις τιμές μέτρησης η υπερβολική νητρορύπανση. Στην, ε, στην νέα νομική πράξη που τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία προβλέπεται πλέον αυτό. Αλλά ακόμα στοιχεία δεν μπορούμε να έχουμε, ακριβώς γιατί δεν έχουν περάσει δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα τέλη της φετινής χρονιάς ή από του χρόνου. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Πέτερ. Ναι, θα μπορούσαμε και να μαλώσουμε αν θέλετε. Δύο χρόνια, λέει ο συνάδελφος, Εξαρτάται όμως από το βάθος των υπογείων υδάτων. Κάποιες φορές χρειάζονται 10 και 15 χρόνια ε, έως ότου εμφανιστούν έως ότου εμφανιστεί η νητρορύπανση στις τιμές μέτρησης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι με ορθολογικό τρόπο παρουσιάστηκε ε, η κατάσταση από την Επιτροπή. Το 2012 έπρεπε να είχε εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Τώρα για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό, δεν το γνωρίζω. Υπήρχαν διαμάχες μεταξύ ε, Υπουργείων ε, και ε, η συνέπεια αυτού ήταν να μην υπάρχει απόφαση. Το 2017 ήταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, τέθηκε σε ισχύ αυτή, αυτός ο νέος κανονισμός της Γερμανίας για τα λοιπάσματα. Φυσικά, ε, μέχρι, μέχρι εκείνη την ώρα, ε, βεβαίω μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, είχαν ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες, επί παραβάση από την Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, το θετικό είναι, όπως είπε και η Κομισιόν, ότι θα το ελέγξουμε ε, και το νέο νόμο της Γερμανίας Και στόχος μας δεν είναι να ελέγξουμε απευθείας αν ε, ε, βελτιώθηκαν οι τιμές, αλλά κυρίως να διαπιστώσουμε αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί ε, κατατείνουν προς τη βελτίωση της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Τι να σας πω, Γερμανός είμαι, φαντάζομαι ότι ο νόμος που αποφάσισε και θέσπισε το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα είναι κατάλληλος για την ε, Γερμανία και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Ελπίζω να γίνει αυτό η ευκαιρία μας επιτέλους να κλείσουμε αυτό το μελανό κεφάλαιο ε, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά θα πρότεινα να παραμείνει ανοιχτή, ανοιχτή η, αναφορία, ε, η αναφορά αυτή μέχρι να πάρουμε και τις τελευταίες πληροφορίες από την Κομισιόν 2012 έως 2017, ε, πέντε χρόνια νομίζω μου είπαν στο σχολείο ότι είναι αυτά. Πολλά μου φαίνονται για να χρειάζεται μια χώρα όπως η Γερμανία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο μια ευρωπαϊκή οδηγία. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, λέει ο πρόεδρος, πράγματι αργοπόρησε η Γερμανία όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στην ε, εθνική νομοθεσία της και αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό ε, πρόβλημα διότι πραγματικά τα νητρικά άλατα είναι ε, εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για την, για υγεία του ανθρώπου. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ενεργή της στάση, τη δραστήρια στάση της. Νομίζω ότι πλέον οδεύουμε προς μια φάση όπου θα μπορέσουμε να κλείσουμε την αναφορά. Δεν έχει έρθει όμως η, η χρονική αυτή στιγμή. Συμφωνώ με τον Πέτερ να την κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Ίσως στην επόμενη συνεδρίασή μας θα μπορούσαμε να επανέλθουμε γρήγορα σε αυτή την αναφορά και να έχουμε ήδη λάβει κάποια θετικά αποτελέσματα. Κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα ε, και ε, να την κλείσουμε πια την ε, αναφορά αυτή. Η επόμενη αναφορά που θέλουμε να επεξεργαστούμε τώρα είναι το σημείο 27 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την αναφορά 11-17 του 2015 που υπέβαλε ο δόκτωρ Φραντσέσκο Ντάτι σχετικά με τον αντίκτυπο ενός ευρωπαϊκού κορονισμού ε, στον πληθυσμό των ρακούν στη Γερμανία. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ μαζί μας, όμως ε, μας παρακολουθεί από το ίντερνετ. Ο Σπύρος Φλεβάρης εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα είδος που εκτίθεται τη ανθρώπινης παρέμβασης έχει βρεθεί εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος με μεγάλο αντίκτυπο στην ε, ποικιλομορφία. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία παρέχει μια λίστα ε, από είδη τα οποία απειλούνται και αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δράσουν με έναν νέο τρόπο για να αντιμετωπίσουν την απειλή στην βιοπικιλότητα. Στη λίστα αυτή βρίσκονται και τα ρακούν και ο αναφέρον ζητάει την αφαίρεση του είδους αυτού από τον κατάλογο ή εναλλακτικά να, τον, να αφαιρεθεί μόνο για τη Γερμανία από τον κατάλογο η, ο κατάρχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά όλα τα κρατημέρια, αλλά άρα αυτό δεν ε, προβλέπεται. Τα επιχείρηματα που προβάλλει ο αναφέρον για την ε, αφαίρεση από την Ευρωπαϊκή αυτή λίστα, από τον κατάλογο, ακολουθούν ε, δύο άξονες. Πρώτον, λένε ότι δεν... ότι θα πρέπει να βρίσκονται στην, στον κατάλογο και αυτή παραμένει η θέση της Επιτροπής, είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ώστε να ε, διωθεί περισσότερο αυτό το είδος γιατί η κατάσταση ο λόγος Ε, που συμπεριλαμβάνεται κάτι σε ένα καταλόγο δεν έχει να κάνει με την κατάσταση τη μεμονωμένη σε ένα κράτο μέλο. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη όπου ταρακούν, έχουν πολύ περιορισμένο. Ε, πολύ περιορισμένη παρουσία και είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η συνεργασία για να αποφύγουμε τον αντίκτυπο, το μελλοντικό που μπορεί να έχει το είδος σε κράτη-μέλη όπου δεν είναι παρόντα. Επίσης, ο αναφέρον συμπεριλαμβάνει και άλλα επιχειρήματα σχετικά με την ευζοία για το είδος και την ε, παρουσία του στον κατάλογο αυτό στο υλικό που μας παρουσίασε περιλαμβάνει πολλά για την εφαρμογή των μέτρων στην Γερμανία, ε, τον κυνηγητικό νόμο, αν αυτό το είδος θα πρέπει να αποτελεί θύραμα, αν θα πρέπει να έχει μια περίοδο προστασίας κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα εθνικής αρμοδιότητες και η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει από αυτού. Αυτό είναι σύμφωνο με τον κανονισμό. Η κατάσταση έχει εξή. Είναι πολύ δεδομένα τα ρακούν στη Γερμανία και ο κανονισμός θεωρεί ότι η Εθνική Αρχή είναι αρμόδια να αποφασίσει τα πιο κατάλληλα μέτρα. Οι ομοσπονδιακές αρχές εγκαίρως κατάφεραν να λάβουν μέτρα διαχείρισης. Θεωρώ τώρα ότι ο διάλογος θα πρέπει να εστιάσει στο πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην Γερμανία όμως δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει το αν θα πρέπει ε, το είδος αυτό να παραμείνει στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Φλεβάρη. Θα ήθελε κάποιος ε, εκπρόσωπος του Γερμανικού Κοινοβουλίου να λάβει το λόγο, ενδεχομένως. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Γιάρ. Μπορεί να θέλουν να τοποθετηθούν και μετά από εμένα. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον κανονισμό για τα χαρακτηριστικά ξένα είδη. Προβλέπεται και μια ευρωπαϊκή διαδικασία για το ποιο μπαίνει στον κατάλογο και ποιο όχι, που δεν εξετάζει πια ε, είδη είναι όμορφα ή λιγότερο όμορφα το κριτήριο είναι αν θέτουν σε κίνδυνο τη βιολογική ισορροπία. Υπήρξαν και διάφορες εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με αυτό το θέμα και το ρακούν για μένα είναι δεδομένο ότι είναι χαρακτηριστικό είδος που θέτει σε κίνδυνο την ε, βιοϊσορροπία ε, στο περιβάλλον της Γερμανίας. Όποιος μάλιστα έχει ε, την παραμικρή ιδέα ε, για περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι πράγματι ε, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα το ρακούν. Αν δεν τεθεί υπό έλεγχο όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή υπό έλεγχο πληθυσμός των ρακούν. Θεωρώ ότι το ρακούν πρέπει να παραμείνει στην λίστα που προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομισμό και θα πρότεινα να κλείσουμε τη συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστούμε, Πέτερ. Την ίδια άποψη συμμερίζονται και οι εμπειρογνωμονές μας και εκείνοι θεωρούν ότι ε, πρέπει να αποδεχθούμε την ε, επιχειρηματολογία της Κομισιόν και να απορρίψουμε τη συγκεκριμένη αναφορά. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής της διάταξης. Θα εξετάσουμε δύο αναφορές. Αφορούν τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους της Γερμανίας. Αφενός έχουμε την ε, αναφορά της κυρίας Αναρίτα Αμορόζο και την αναφορά του κυρίου Καρλ Χέρ. Σχετικά με ε, τα διόδια στη Γερμανία. Και τους ε, Γερμανούς υπηκόους που ζουν στο εξωτερικό. Αναρίτα Αμαρόζου, είστε εδώ. Έχετε το λόγο. Γεια σας. Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι ε, εκπρόσωποι της Bundestag, τον Οκτώβριο η Αυστρία στις 12 Οκτωβρίου έστειλε στην Γερμανία μια κλήτευση που αφορούσε την παραβίαση του 1834 και του 1992. Αυτά τα τρία άρθρα όσον αφορά τη λειτουργία της ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αυτές οι διατάξεις ε, αφορούν τα τέλη όσον αφορά τις μεταφορές. Και όλοι όσοι χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους στη Γερμανία πρέπει να πληρώσουν κάτι σαν διόδια για τις υποδομές επί τη βάση των εκπομπών του αυτοκινήτου που οδηγούν. Και όσοι μένουν στη Γερμανία μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω υπό τη μορφή κάποιες φοροαπαλλαγής. Οπότε έτσι τελικά επιβαρύνονται μόνο οι αλλοδαποί οι οποίοι οδηγούν στο κινητοδρόμους. Επομένως αυτό είναι δυσμενής έμεση διάκριση. Και έτσι παραβιάζεται το άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η άνηση μεταχείριση αφορά το ότι ο έλεγχος αυτής της επιβάρυνσης για το αν έχουν υποβληθεί ή όχι αυτά τα τέλη, αυτό θα εφαρμοστεί μόνο όσον αφορά τους ξένους οδηγούς. και όχι όσον αφορά τους Γερμανούς. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως να θέσει στο αργείο τη σχετική καταγγελία. Άρα χρειάζεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατόπιν της συμφωνίας του Παρισιού ε, πρέπει η διεθνής κοινότητα να κινηθεί προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια κινητικότητα καθαρή από τέτοιες εκπομπές. Οπότε θα πρέπει και η βιομηχανία μας αντίστοιχα να γίνει πρωτοπόρα με καινοτομία και ψηφιακά, να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε Κίνα και ΙΠΑ. Έτσι, η ψηφιακή τεχνολογία θα κάνει πιο ευφυή και πιο αποτελεσματική την κινητικότητα, ούτω ώστε αυτό να καλύψει και τις μεταφορές και να υπάρχει διαφοροποιημένη χρέωση των διοδίων και η χρέωση να γίνεται με κάποιο είδου ε, τηλεχειριστήριο. Οπότε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ψηφιακή τεχνολογία. Τον Ιούνιο η Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την οδηγία αυτήν για να υπάρχει διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Θεωρήθηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σχετική νομοθεσία και τα κρατημέλη και οι γειτονιάρουσες χώρες έτσι θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και έτσι θα επιτευθούν οι στόχοι της πολιτικής μεταφορών. Άρα δεν θα χρειάζονται πλέον αυτές οι βινιέτες με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Άρα χρειάζεται ένας κανονισμός που να επιτρέπει την ανταλλαγή των πληροφοριών μέσω νομικών συμφωνιών και έτσι τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται. Επί τη βάση όλων αυτών των επιχειρημάτων θέλω να μείνει η αναφορά ανοιχτή έως ότου αποφασίσει και κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ε, αυτός ο νόμος ο γερμανικός που θα με το 19 να μην ισχύει κατά αυτό τον τρόπο να μην υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση βάση εθνικότητας. Χρειάζεται να εφαρμόσει τη αρχή της ε, αλληλεγγύης μεταξύ των ε, πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φρέντρικ Ρασμούσεν, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μας παρουσιάσει την επίσημη θέση της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, να σας πενθυμίσω ότι από πλευρά κοινωνική νομοθεσία δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση για επιβατικά, αλλά μόνο για μεγάλα φορτηγά. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τη Γερμανία 28 Ιουνίου όσον αφορά το νομοσχέδιο για την επιβάρυνση αυτών των ε, οχημάτων θεωρήθηκε για τα λοδαπά οχήματα δυσμενής διάκριση. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο επέλεξε να τροποποιήσει την πρώτη πρόταση, να λάβει υπόψη τι είπε η Κομισιόν σε σχέση με τη διαδικασία η παραβάση. Κατόπιν θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει πλέον περίπτωση δυσμενής διάκρισης διότι η συσχέτιση οχήματος και ε, χρέωσης και δυο-δύο αν θέλετε δεν υπήρχε πλέον. Οπότε υπήρξε αυτή η πρόταση για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά αυτά τα μεγάλα φορτηγά και προβλέπεται Τώρα η συμπερίληψη των επιβατηγών. Η πρότασή μας αποσκοπεί στο να γίνεται η χρέωση βάσει απόστασης διανυόμενης. Όλοι να πληρώνουν τα ίδια για να μην υπάρχει δυσμενής διάκριση. Τα ίδια ανά χιλιόμετρο που διανύουν. Αυστρία στη συνέχεια αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυνάμει το 259 της ε, συνθήκης. Κυρίως γιατί διαφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από δικής μας πλευράς έχει εκφύγει τον γύρο μας η υπόθεση, έχει κλείσει η υπόθεση για μας και τώρα από τις 13 Οκτωβρίου του 2017 έχει επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε έναν χρόνο αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εμείς συστήνουμε να κλείσει η αναφορά αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Ράσμουσεν. Κύριε Γιάρ, πρότεινε να αλλάξουμε τη σειρά των τοποθετήσεων. Θα ήθελε κάποιος ευρωβουλευτής λοιπόν να τοποθετηθεί, ίσως εσύ ο ίδιος. Ναι, κάτι έχω να πω κι εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μια γενική πολιτική εκτίμηση να εκφράσω. Η εναρμόνιση των διοδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι η χειρότερη δυνατή ιδέα. Γιατί ε, ε, αν κάθε ένας ε, δημιουργεί το δικό του σύστημα Εντάξει, τα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, πηγαίνουμε και στο Στρασβούργο. Ήδη έχουμε ένα αυτοκόλλητο, μια βινιέτα για το, για την... για το Στρασβούργο. Μου έχει τύχει όμως να βρεθώ και με αυτοκίνητο στην, στην Πορτογαλία, όπου δεν είχα το αντίστοιχο αυτοκολλητάκι στο παρμπρίζ μου. Στο τέλος θα γεμίσουν τα παρμπρίζ μας αυτοκόλλητα. Ε, οπότε θα έλεγα ότι να γίνει ένας απολογισμός και να κινηθούμε προς μία κάποια εναρμόνιση. Ώστε να μπορεί κανεί να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρί να χρειάζεται κάθε φορά που περνά τα σύνορα να, να, να κολλάει και να ξεκολλάει αυτοκολλητάκια από το παρεμπρέις του. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά αυτά δεν θα ε, διευθετηθούν σε λί... Ε, από τη μία μέρα στην άλλη. Χρόνια θα χρειαστούν να συζητήσουν, αλλά μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο διάλογο, γιατί όχι. Ε, δεν μπορούμε όμω σε κάθε περίπτωση να έχουμε ενιαία αγορά χωρί δασμού κτλ, κτλ. Αλλά να μην μπορεί κανεί να περάσει από τη μία χώρα στην άλλη ε, με το αυτοκίνητό του. Το δεύτερο θέμα είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο. Η Κομισιόν τα παρουσίασε με εξαιρετικό τρόπο. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Το 2015 είχαμε μια καταγγελία, την έλαβε πίσω. Στη συνέχεια ε, λάβαμε μια νέα εκδοχή όπου η Κομισιόν μας είπε ότι δεν είναι διακριτική μεταχείριση αυτό που συμβαίνει είναι όμως ε, τμήμα της ε, δημοκρατικής ένομης τάξης αν θέλετε να μπορεί κάποια χώρα που διαφωνεί με μια απόφαση της Κομισιόν να προσφύγει στο δικαστήριο. Περιμένουμε λοιπόν τι θα αποφανθεί το δικαστήριο να δούμε Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε την αναφορά και να την αφήσουμε ανοιχτή και να την ε, ε, κλείσουμε. Δεν θα επιμείνω όμω ούτε στη μία άποψη ούτε στην άλλη. Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να την ε, κλείσουμε. Για να πάρουμε μια απόφαση. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση γιατί εκτιμώ πολύ το, το σύστημα των αυτοκινητοδρόμων στην Γερμανία και λαμβάνει υπόψη τα ε, συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Τώρα να πάρει το λόγο εκπρόσωπο ε, τη γερμανική βουλή. Θα μιλήσω για το δικό μου κόμμα. Στη Γερμανία. Είναι, η Γερμανία είναι χώρα διέλευση στην Ευρώπη. Έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό δικό δίκτυο. Το 15% της κυκλοφορίας δεν είναι Γερμανοί καθώς είμαστε χώρα διέλευσης, έχουμε ανοιχτά σύνορα και αυτό το σύστημα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρηματοδοτούμε, θα πρέπει να τις επεκτείνουμε, ε, να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Εμείς ως κόμματα προτείνουμε να εισάγουμε ένα ε, διόδια της άξης των 80 ευρώ για τα βαρέα οχήματα ετησίως. Σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν χαμηλότερο ε, ποσό ορισμένο στην ε, είναι 3 με 5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα 7,8 το είναι το ετήσιο ποσό στην Ελβετία. Είναι σημαντικό για αυτό για μας, αλλά παράλληλα προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, ε, να δούμε την πρωτοβουλία να υπάρξει συναρμόνιση. Αυτό που είπε ο Σανθός Γιάρ, ότι σε κάθε σύνορο, σε όλα τα σύνορα χρειαζόμαστε ένα καινούριο αυτοκόλλητο, Και φυσικά είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς είμαστε, λειτουργούμε ανεξάρτητα από τα διόδια που έχουν επιβληθεί και έχουμε προσαρμόσει και την νομοθεσία την περιβαλλοντική για να υποστήριξουμε την περιβαλλοντική διάσταση. Αυτός είναι και ο σκοπός σας εδώ, στο πλαίσιο της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για να καταργήσουμε και τα παλιά πετρελαιοκίνητα οχήματα. Άρα, είμαστε υπέρ Ε, του γεγονότο ότι ε, δεν υποστηρίζεται και από την Επιτροπή αυτή, αυτό το αίτημα και ότι θα πρέπει να κλείσει. Λοιπόν, η εναρμόνωση εντός της Ευρώπης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά συστήματα θα έχουμε αν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Έκανα μια μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι για να δούμε πόσα αυτοκόλλητα μπορεί να μαζέψει κανείς στο παρμπρίστου. του. Θεωρώ όμως ότι είναι και μια σημαντική υπόφαση όταν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία η παραβάση Θεωρούμε ως κομμό ότι είναι δύσκολο μια τέτοια αναφορά σε ένα τέτοιο σημείο να την, να, την κλείσουμε. Οπότε διαφωνώ με τους συναδέλφους μου. Έχω όμω την αίσθηση ότι όταν υπάρχει, όταν ε, τρέχει μια διαδικασία δικαστική, δεν μπορούμε προτού βγει η απόφαση να κλείσουμε την σχετική αναφορά. περιμένουμε τις ε, αποφάσεις τις δικαστικές πρώτα και μετά καθορίζουμε τις αποφάσεις μας. Στη Γενική Βουλή είχαμε μία αναφορά πρόσφατα που είχε να κάνει Da haben wir die unterschiedlichsten Systeme innerhalb την επιβάρυνση σωματιδίων που προκύπτει από τα βαρέα οχήματα. Θα ήταν λοιπόν σωστό να δούμε μια εναρμόνιση και σε αυτόν τον τομέα. Όταν κάποιο ε, περνάει από περισσότερες ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να έχει και τα κατά τις κατάλληλες πλακέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ οι φιλελεύθεροι στο Γερμανικό Κοινοβούλιο έχουν ελαφρώς διαφορετική άποψη. Για να σας δώσω κάποιους αριθμούς. Ε, τα τέλη κυκλοφορίας ε, ανέρχονται σε 50 δισεκατομμύρια ε, στη Γερμανία. Η, τα έξοδα μας, οι δαπάνες μας ανέρχονται σε 34 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Γενικά δηλαδή εισπράττουμε αρκετά χρήματα από τέλη κυκλοφορίας. Απλά δαπανώνται ε, με σφαλμένο τρόπο. Είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Και θεωρούμε ότι έχουμε πλέον μια σχεδόν ολοκληρωμένη ε, οικονομική ένωση. Έχουμε νομισματική ένωση, τα, τα, τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη, το ίδιο και τα προϊόντα, τα εμπορεύματα. Οι εργαζόμενοι της ε, Ευρώπης μπορούν να εγκαθίστανται και να εργάζονται όπου θέλουν, αλλά τα αυτοκίνητα για κάποιον λόγο πρέπει να τα χειριζόμαστε διαφορετικά. Ε, διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να καθοριστεί ε, ευρωπαϊκό ε, σύστημα διοδίων. Αντίθετα, θα θέλαμε να καταργηθούν παντού. Επίσης, γνωρίζουμε στην Γερμανία ότι τα διοικητικά έξοδα που συνοδεύουν ε, την, τα διόδια θα είναι είτε ίσα είτε και μεγαλύτερα από τα έσοδα που θα αποφέρει η εισαγωγή ενός συστήματος διοδίων. Γι' αυτό και απορρίπτουμε συνολικά ε, τα διόδια. Πρόεδρος, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Εκ μέρους του Τσέσου στον Bundestag θέλω να τοποθετηθώ πολύ σύντομα και πολύ γενικά. Ε, όσο βρίσκεται ε, υπό εξέταση η υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε την απόφαση που θα, στην οποία θα καταλήξει το δικαστήριο. Έχουμε τις αναφορές βεβαίως για να μην ξεχαστεί το θέμα. Ε, εγώ λοιπόν ε, θα πρότεινα να κλείσετε την ε, υπόθεση αυτή και να επανέλθουμε στην υπόθεση αυτή όταν πια θα έχουμε στα χέρια μας και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Πέτερ. Ναι, βλέπετε κύριε Πρόεδρε, μόλις μιλάμε για αυτοκίνητα, ξαφνικά ξυπνάει η γερμανική ψυχή από το λίθαργο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό και στους συντονιστές και να το, ε, ε, να το συζητήσουμε και μεταξύ των πολιτικών ομάδων, γιατί δεν είναι όλες εδώ και σε αυτή την περίπτωση βλέπω ότι υπάρχουν καλά επιχειρήματα και από τι δύο πλευρέ και εν πάση περιπτώσει με επιβεβαίωσαν σε αυτή την άποψή μου και οι συνάδελφοι από, τον, από, το, από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ε, ο, πάντως, ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Μπορείτε να την κλείσετε, μπορείτε να αφήσετε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή. Εγώ ό,τι και να αποφασίσετε θα σας στηρίξω. Πρόεδρος, ωραία, πρωτού αποφασίσω για το τι θα κάνουμε με την αναφορά αυτή θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην αναφέρουσα ε, για μια τελευταία φορά. Παρακαλώ. Ε, με άπειρη ικανοποίηση διαπιστώνω όλα αυτά που είπαν οι κύριοι πριν ε, ε στα γιατί πάνω ότι αποδέχονται την κρίση του δικαστηρίου και ότι οι συνέπειες αυτής της απόφασης έχουν σχέση με την αναφορά Οπότε ε, βεβαίω θέλω να μείνει ανοιχτή. Και βλέπω ότι και άλλοι έχουν ζητήσει την ίδια διαδρομή. Και άκουσα τον κύριο Ούλρικ και εγώ θέλω να καταργηθούν τα διόδια. Εδώ να υπάρχει κάποια ενεργοσμένη ρυθμίση σε όλη την Ευρώπη και στην Ιταλία άλλωστε πληρώνουμε πάρα πολλά. Ε, έχουμε όλες αυτές τις ε, ε, κουραστικές ε, αυτοστράντες ε, δεν είναι και καλύτερε οι προσφέρομενες υπηρεσίες οπότε θα ε, έπρεπε να επιληφθεί η Ευρώπη να εναρμονίσει το θέμα για όλα τα μέλη της Ένωσης ενδεχομένω θα μπορούσε στην επόμενη θητεία να θεωρηθεί η υπόθεση μια προτεραιότητα για μένα αυτό αποτελεί νίκη θρίαμβο ευχαριστούμε. Λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξή. Αναμφίβολα έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που προκαλεί πολλές διαφωνίες και διχογνωμίες. Θεωρώ ότι η Κομισιόν επίση περιέγραψε με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο την κατάσταση. Γεγονό είναι ότι αυτή τη στιγμή εκρεμεί η υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυρία Μορόζο, θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Αναφορών έφτασε στα όρια της. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Ε, το πράγμα πλέον το επεξεργάζονται εκείνοι που ε, είναι αρμόδιοι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δηλαδή. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που μας είπατε και αυτά που μας είπαν όλοι οι παρόντες και θα πρότεινα να κλείσουμε την αναφορά αυτή, ακόμη και αν διαφωνείτε. Δυστυχώ έτσι και αλλιώ δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα όσο το θέμα εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μετά την απόφαση ε, αν δεν σας ικανοποιήσει η απόφαση, ε, τότε βεβαίως θα έχετε και πάλι το δικαίωμα να υποβάλλετε νέα αναφορά, την οποία βεβαίως και θα επεξεργαστούμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Ακούσαμε επίσης πάρα πολύ καλές προτάσεις. Ενδεχομένως ε, τελικά να επιλεγεί και μια πανευρωπαϊκή εναρμόνιση των συστημάτων διοδίων. Ε, και νομίζω μπορεί και να, μην, ε, να κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι σας ικανοποιεί και αυτή η απόφασή μου, αυτή η εξήγηση που σας έδωσα και όπως είπα μόλις βγει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ο κύριος Στέφαν Βάχτλερ υπέβαλε αναφορά υπαριθμών 0879 σχετικά με την παρουσία, ε, την θέσπιση κανονισμού στη Γερμανία ε, ε, που διέπει τα τρανς λιπαρά οξέα στα τρόφιμα. Έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος και θα έχει το λόγο τώρα για να μας παρουσιάσει τη θέση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα σήμερα είναι η κατανάλωση τρανς λιπαρών οξέων που ε, ε, ενισχύει τις ε, ασθένειες του κυκλοφορικού μέσω της αύξησης της χολυστερίνης. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και έχει επιβεβαιωθεί και από, την, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων. Σε μια σειρά από χώρες, όπως για παράδειγμα τη Δανία έχουν θεσπιστεί ε, νόμοι ε, για τον περιορισμό της περιεκτικότητας των τροφίμων σε τρανς λιπαρά. 2% συγκεκριμένα είναι το όριο που ορίζεται στην νομοθεσία της Δανίας. Η Κομισιόν εξετάζει το θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Βάσει ετοιμάτων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε στα τέλη του 2015 μια πρώτη έκθεση όπου Εξετάστηκε η περιεκτικότητα των τροφίμων σε τρανς λιπαρά οξέα στα διάφορα κράτη-μέλη και εξετάστηκαν διάφορες επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εξετάσαμε γιατί αν θα έπρεπε να επισημένονται τα τρόφιμα αυτά ή αν θα ήταν καλύτερη επιλογή να προβούμε σε περιορισμό της ε, επιτρεπτής περιεκτικότητας. Στη βάση λοιπόν της έκθεσης εκείνη εκπονήθηκε και μια περαιτέρω μελέτη που επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο που θα είχαν οι διάφορες δυνητικές επιλογές στην οικονομία, στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2017, η οποία και ελήφθη υπόψη σε μια μελέτη αντικτύπου, η οποία παρουσιάστηκε στα μέσα του 2018. Και το αποτέλεσμα αυτής της πολιετούς διαδικασίας μπορώ με χαρά να ενημερώσω τον κύριο Βάχτλερ ότι πλέον υπάρχει ε, σχέδιο νομικής πράξης η οποία και παρουσιάστηκε στις 4 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα σχέδια νομικών πράξεων δημοσιεύονται ε, για τέσσερις εβδομάδες ε, και στη διάρκεια αυτή μπορεί κανείς, ε, ο, οποιοδήποτε πολίτες, ο πολίτης να υποβάλει σχόλια. Βεβαίως κοινοποιήθηκε το σχέδιο αυτό της νομικής πράξης και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και για δύο μήνες τα κράτη-μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο κανονισμού. Περιορισμός ε, των ε, ε, τρανσλιπαρών για βιομηχανικά προϊόντα και εδώ επίσης χρησιμοποιήσαμε αυτό το 2% της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά για τον τελικό καταναλωτή το αντιστοιχεί, όπως είπα, και σε αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται στην νομοθεσία και ευρωπαϊκών αλλά και μη ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ αυτών και στην νομοθεσία της Δανίας. Αυτά από πλευράς μας, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και βεβαίως στη βάση της αναφοράς σας ε, βεβαίως θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διαβιβάσουμε σε εσά όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Πέταγια όσον αφορά το περιεχόμενο και αν καταλαβαίνω καλά την αναφορά αυτό που είναι επιθυμητό είναι νομοθετική ρύθμιση οπότε προτείνω να κλείσουμε την αναφορά εφόσον προβλέπετε κάτι τέτοιο γιατί ουσιαστικά έχει εκπληρωθεί το αίτημα Πιστεύω ότι η είδηση αυτή από την Επιτροπή ήταν πολύ καλή για τον αναφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Πέταγιά μόλις τώρα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που μας παρουσιάσετε ο αναφέρον θέλει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει τα πρώτα, έχει κάνει τα πρώτα βήματα για το πώ θα είναι αυτός ο κανονισμός. Θεωρώ όμως ότι έχει εκπληρωθεί το αίτημα του αναφέροντα, άρα μπορούμε να την κλείσουμε. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις μπορούμε να την κλείσουμε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 31 της ημερήσιας διάταξης «0963» έχει για την αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων ε, στον υγειονομικό κλάδο. Από όσο γνωρίζω, είναι παρόν ο αναφέρον, είναι στην αίθουσα. Ο λόγος εσάς κύριε Χουσάνο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο αναφέρον. Κύριε Βουλευτέ, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ σήμερα και να μιλήσω για λογαριασμό περίπου 100.000 νοσοκόμων από Βουκουρέστη και γενικότερα από την ε, Ρουμανία. Αυτό το οποίο θέλουμε την αναφορά είναι να αναδείξουμε ε, τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι νοσοκόμοι στη χώρα μα. Ε, σήμερα στην ε, Ρουμανία έχουμε νοσοκόμους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά αλλά έχουν μεταξύ τους ανισότητα μισθολογική γιατί ο μισθός στηρίζεται ε, στην παιδεία που έχουν λάβει, στους τίτλους σπουδών που έχουν. Μπορούν να σπουδάσουν σε διάφορα μέρη, σε σχολές, σε πανεπιστήμια, σε τεχνικές σχολές, σε ε, διάφορα ιδρύματα που είναι μείγμα τεχνικής σχολής και πανεπιστημίου κλπ. Οπότε έχουν διαφορετικές επιλογές μπροστά τους. Και υπάρχει επίσης ε, ένας τίτλος σπουδών που ανησυχεί στο ίσκε 2 και ένα άλλο που ανησυχεί στο ίσκε 3. Το σχετικό νόμος τροποποιήθηκε το 2017 και θεσπίστηκε ένα μηχανισμό για την μετατροπή των ε, τίτλων σπουδών προσαρμογή στα σημερινά. Όμως δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ιδρύματα προς να κάνουν αυτό που λέει ο και επομένω πολύ λίγοι μπορούν να κάνουν αυτή τη μετατροπή. Οπότε έχουμε ε, περίπου 100 μόνο νοσοκόμους από όλη την χώρα και νοσοκόμες που το έχουν κάνει, έχουν κάνει αυτή την ε, προσαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι ε, αν 100 μπορούν κάθε χρόνο να κάνουν αυτό που πρέπει, σημαίνει ότι χρειάζονται χίλια χρόνια για να καλυφθούν όλοι οι νοσοκόμοι. Οπότε έχουμε τέσσερα χρόνια προπτυχιακά τώρα που περνούν οι νοσοκόμοι και οπότε θέλουμε να μας βοηθήσετε όσον αφορά την τυποποίηση των σπουδών για τους ε, μελλοντικού νοσοκόμους και νοσοκόμες ούτως ώστε όλοι να έχουν την ίδια κατάρτιση εκπαίδευση. Επίσης θέλουμε να βοηθήσετε ούτως ώστε να υπάρξει ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ε, κατάρτισης και έτσι να αναβαθμίζονται και να προσαρμόζονται στα ισχύοντα οι σπουδές των νοσοκόμων. Οι δικαιούχοι επομένως μπορούν να αναβαθμίζουν ε, τη προσόντα τους, τις δεξιότητές τους, Αυτά τα έχει κάνει επιτυχώ και η Ισπανία και το Βέλγιο. Οπότε είναι και θέμα μισθολογικό. Θα είχαμε σε περίπτωση που τα καταφέρναμε μια ισότητα. έχουμε κάποιες ε, οδηγίες που απαιτούν το να υπάρχουν αντισταθμίσεις στα θέματα της ε, επαγγελματική κατάρτισης πριν από κάποια χρόνια υπήρξε η ευκαιρία πλευράς δικαίου για την αναβάθμιση των ε, δεξιοτήτων και τίτλων σπουδών. Όμως αυτό περιορίστηκε στο πώς θα μπορέσουν οι Ρουμάνοι να δουλέψουν σε άλλα κρατημέλη. Δεν λύθηκε το πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε και άλλες μορφές δυσμενούς διάκρισης. Νοσοκόμοι, νοσοκόμες με καλύτερους τίτλους σπουδών, καλύτερες δεξιότητες, υφίστανται δυσμένη διάκριση και θα έπρεπε να πληρώνονται περισσότερο. Έχουμε 28.000 Ρωμανούς που έχουν φύγει και έχουν πάει αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι έχουμε αυτό το διπλό σύστημα το οποίο θα έπρεπε να καταργηθεί και να υπάρχει ενιαία κατάρτιση και εκπαίδευση. Γι' αυτό και προσφυγούμε σε αναφορά. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χασάν. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Επιτροπής. Ο κύριος Τομάρας, δεν είμαι σίγουρος ποιος από τους δύο θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος. Το γνωρίζαμε μόνο από τα έγγραφα. Πρώτα-πρώτα. Για να δούμε λίγο το πλαίσιο. Τι γίνεται με την ε, οργάνωση της υπηρεσίας, τι γίνεται με την πολιτική υγεία, τι γίνεται με τις ε, ιατρικές υπηρεσίες που είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Έχουμε βέβαια κάποιες εξαιρεσει και μία από αυτές είναι η ελάχιστη εναρμόνιση που θα πρέπει να έχει γίνει για το τι θα ρυθμίζουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τους νοσοκόπους. Αυτές οι ελάχιστες ε, με την τροποποίηση και τις οδηγίας τροποποιήθηκαν το 2013. Όσον αφορά δηλαδή τη διάρκεια ε, της, ε, ε, της κατάτησης, τρία χρόνια, 4.600 ώρες και θα πρέπει ο κάθε νοσοκόμος νοσοκόμα καθορίζει τι πρέπει να μεταίνει. Αυτό είναι το ελάχιστο. Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να ανεβάσουν τον πύχη πέραν αυτού του ελαχίστου ή μπορεί να αποφασίσουν να περιοριστούν σε αυτό το προβλεπόμενο ελάχιστο. Σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι να υπάρχει δηλαδή ομοιομορφία σε ενεργο επίπεδο, η οδηγία είναι δύο δυνατότητες στα κρατη μηλη Πανεπιστημιακή κατάρτιση ή επαγγελματική κατάρτιση. Και από εκεί το κράτος μέλος να επιλέξει. Ίσως ο κράτος μέλος διαλέξει και τα δύο επίπεδα. Ίσως το κρατός μέλος μπορεί να θέλει δύο διαφορετικούς τρόπους κατάρτισης. Όλα αυτά συμβαδίζουν με το κοινωτικό δίκαιο. Αλλά πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα όσον αφορά το περιεχόμενο, τη διάρκεια κλπ. Όποια έτσι οι αρχές της χώρας, αν θέλουν, μπορούν να έχουν μόνο τον ένα κλάδο, δηλαδή ας πούμε πανεπιστημιακή κατάρτιση, αλλά δεν υποχρεούνται. Έγινε αυτή η τροπήση το 2017 και όλα θα πρέπει τώρα να συμμετέχουμε την οδηγία. Πάλι υπήρχαν περισσότερες επιλογές, τώρα υπάρχουν αυτές που είπαμε. Οπότε υπάρχουν τώρα στην αγορά κάποιοι επαγγελματίε νοσοκόμοι που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το παλιό καθεστώ. Από πλευρά τώρα ελεύθερη διακίνηση έχουμε διαφορετικού κανόνε αναγνώριση των δεξιοτήτων να μπουν στο εξωτερικό όπω και εσεί είπατε. Άρα θα υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι αναγνώριση. Αυτοί επομένω που τηρούν τι ελάχιστε προδιαγραφέ έχουμε αναγνώριση αυτόματη. Όσοι όμως ακολούθησαν άλλο τρόπο κατάρτισης αυτοί θα πρέπει να απαντήσουν, σίγουρα να αποδείξουν ε, χρόνια εμπειρίας, πρακτική εξάσκηση για να μπορούν να δουλέψουν σε άλλο κράτος μέλος. Όπως προαναφέραμε, είναι θέμα ελεύθερης διακίνησης. Όλα αυτά επομένως αφορούν τη διασυνοριακή μετακίνηση των νοσοκόμων. εσεί θέλετε, όλα αυτά να ισχύσουν και στο εσωτερικό τη χώρας και να έχετε αντισταθμιστικά μέτρα για όσους ε, έκαναν την παλιά εκπαίδευση και να μπορούν να δουλέψουν με τις ίδιε συνθήκε. Αυτό όμως δεν εμπίπτει στην ε, οδηγία. εκεί στη Ρουμανία ε, το πώς θα ρυθμίσει το ιστορικό ε, σύστημα. Όσον αφορά την αμοιβή, δεν λέει τίποτα η οδηγία. Άρα δεν αποκλείει το να συνδέεται ο μισθός με την κατάρτιση. Είναι αρθινική αρμοδιότητα να ρυθμίσει την αμοιβή, το μισθό σε σχέση με το σύστημα κατάρτισης. Ελπίζω ότι σας διαφώτισα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ερώτη προς τους βουλευτές. Θέλει κάποιος το λόγο. Συνάδελφοι, όπως βλέπετε η Ρουμανία αιμορραγεί όσον αφορά το προσωπικό της, τους επαγγελματίες υγείας της ε, προς άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20% των επαγγελματιών έχουν ε, εγκαταλείψει τη χώρα. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στον, ε, στη χώρα μου. Η αναφορά αυτά, αυτή με τις 7.000 και πλέον υπογραφές είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο της υγείας στη Ρουμανία. Για να σταματήσει λοιπόν η διάκριση, η μισθολογική στον ε, κλάδο, πρέπει να αναλυφθεί δράση. Ο κλάδος αυτός ε, έχει διέλθει από διάφορους κανόνες, διάφορα συστήματα οργάνωσης στη Ρουμανία, στην πάροδο των χρόνων και υπάρχει μια διάκριση μεταξύ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι μια διάκριση η οποία δεν υπάρχει σε άλλες ε, χώρες. Θεωρητικά μπορεί κανείς να αναβαθμίσει το πτυχίο του. Στην πράξη όμως δεν, δίνεται, δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα στους Ρουμάνους πολίτες που εργάζονται στον κλάδο της υγείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πανεπιστημιακούς ε, ε, ε, ε πανεπιστημίου με λιγότερη εμπειρία που αμείβονται όμως με υψηλότερους μισθούς από ε, νοσηλευτές που έχουν ε, μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Θα έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάποιες εξετάσεις ή να αναγνωρίζεται τουλάχιστον η εμπειρία τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αποζημίωσης όσον αφορά την ε, επαγγελματική εκπαίδευση σε άλλα κράτη-μέλη. Στην Πολωνία, την Εστονία, το Βέλγιο ε, και την Ισπανία έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Και από, αυτά, από αυτές τις χώρες πρέπει να παραδειγματιστούμε και εμείς. Πρόεδρε, θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το αν η Ρουμανία συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία. Και αυτό δεν αφορά μόνο ε, τους 7.521 που υπέγραψαν την αναφορά, αλλά τους 20.000 νοσηλευτές που εργάζονται στην Ρουμανία. Ο Πέτερ Γιάρ έχει το λόγο. Ε, αντιμετωπίζω πρόβλημα πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε. Αφενός αντιλαμβάνομαι και δέχομαι αυτά που μας λέει ο αναφέρον. Θεωρώ ότι είναι δίκαια τα αιτήματα αυτά και εύλογα. Βεβαίως θα πρέπει κανείς να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετες δεξιότητες αν αυτές απαιτούνται από την νομοθεσία. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να καθορίζουν τα συστήματά του όσον αφορά την παροχή των επιπλέον δεξιοτήτων. Η Κομισιόν, απ' την άλλη, μα λέει ότι όλα αυτά επιτρέπονται, αλλά εναπόκειται στα κράτη-μέλη να τα αποφασίσουν. Κυνηγάμε την ουρά μα δηλαδή. Άρα, αυτό που ζητάει ο αναφέρον επιτρέπεται αφενό από την οδηγία, έτσι μα λέει η Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόσει η Ρουμανία, η οποία όμω δεν τα εφαρμόζει. Εγώ θα πω ξεκάθαρα. Το αίτημα του αναφέροντος είναι δίκαιο. Μπορούμε λοιπόν ως Επιτροπή Αναφορών να αποστείλουμε μια επιστολή στις Ρουμανικές Αρχές όπου θα τις ρωτάμε για ποιο λόγο δεν κάνετε αυτά που μπορείτε να κάνετε γιατί δεν αξιοποιείτε τις αρμοδιότητες σας ε, αυτά που μπορείτε να κάνετε. Το ερώτημα όμως είναι θα το προσεγγίσουμε με αυστηρότητα ή όχι. Αφενό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι δική μα αρμοδιότητα, οπότε κλείνουμε την αναφορά. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι αν την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, τότε θα ασχηθεί πίεση στι ρουμανικέ αρχέ. Γι' αυτό είμαι κάπως διχασμένος. Αφενός θα έλεγα, να, η άποψη μου θα ήταν να κλείσουμε την ε, αναφορά. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω ότι η αναφορά, αν παραμείνει ανοιχτή, ασκείται ποιήση. Αλλά ίσως είναι και πολιτικού χαρακτήρα η απόφαση που θα λάβουμε. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στον αναφέροντα ότι δεν ε, συμφωνούμε με αυτά που κάνει η ρουμανική κυβέρνηση. Δεν έχει πολύ νόημα βέβαια. Δεν δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ ε, εύλογα αυτά που κάνει η ρουμανική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά επιτρέπονται με βάση την, την οδηγία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, συμφωνώ. Ε, με τον Πίτερ συμφωνώ, λοιπόν. Σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε περάσει τη διαδικασία του να έχουμε ισότιμες αμοιβέ σε πολλούς τομείς, ίσες αμοιβέ. έχουν γίνει αλλαγές ε, ρυθμιστικές όσον αφορά τα προσόντα και τις, ε, τα κλιμάκια, τα μισθολογικά. Ίσως στέλνοντας μια επιστολή στις ρουμανικές αρχές, όταν κλείσουμε την αναφορά αυτή, θα μπορούσαμε να τους ενθαρρύνουμε να δουν πώς τα άλλα κράτη-μέλη κατάφεραν, να διασφαλίσουν ε, ίσως μισθούς γιατί πολλοί βρέθηκαν σε πιο δυσχερή θέση κατά αυτής της διαδικασίας. Άρα το θεωρώ χρήσιμο αυτό να υπάρξει σαν κάτι πρόσθετο μαζί με την επιστολή. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί. Παρακαλώ τον αναφέροντα να πάρει το λόγο. Πράγματι, 100.000 νοσηλευτέ νοσηλευτές στην Ρουμανία θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδέ τους. Το κράτος της Ρουμανίας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα το 2017, αλλά ούτε ένα πανεπιστημίο στην Ρουμανία δεν προσφέρει δυνατότητα τέτοια. Αν τα ρουμανικά πανεπιστήμια βοηθούσαν στην μεταφορά ε, μονάδων θα χρειαζόταν ε, πάρα πολλά χρόνια για, τις, για για να μπορέσουν να το πετύχουν αυτό. Είναι κάτι μη ρεαλιστικό και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις δύο προτάσεις. Έναν τρόπο κατάρτισης, μία μέθοδο κατάρτισης και κρατικές εξετάσεις για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους. Αν θα μπορούσα να έχω το λόγο για μερικά ακόμα δευτερόλεπτα. Για να μπορεί κάποιος να εκπαιδεύσει τους νοσηλευτές, πρέπει να είναι ο ίδιος νοσηλευτής. και με την τρέχουσα κατάσταση αυτό χρειάζεται να κάνει κάποιος προπτυχικές σπουδές και μεταπτυχιακές σπουδές και να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, θα κάνω την εξής πρόταση και θα ζητήσω συγγνώμη Η αυστηρή προσέγγιση, νομική προσέγγιση του θέματος. Ε, λοιπόν, έχει ακούσει ο αναφέροντας τις απόψεις μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμόδιότητα σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να πω, γιατί είναι web streamed η συνεδρίασή μας. Περισσότεροι συνάδελφοι, από ό,τι βλέπω, είναι υπέρ του να κλείσουμε την αναφορά. Εγώ όμως διαφωνώ. Θα έλεγα πως ήταν καλύτερο. Είναι και ψυχολογικό το θέμα. Κατανοώ ότι πολλοί στη Ρουμανία, πολλοί πολίτες περιμένουν από εμά να αναλάβουμε δράση από τη στιγμή που δεν κάνει κάτι η ίδια η χώρα τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την αίσθηση ότι σε έχει εγκαταλείψει έχετε αισθάνθει την εγκατάλειψη στην πρώτη, στον πρώτο γύρο των συζητήσεων και αυτό σας έχει επηρεάσει ψυχολογικά. Οπότε αυτό προτείνω είναι να αποστείλουμε μια επιστολή στη ρουμανική κυβέρνηση και σας παρακαλώ να ε, εκφραστείτε επί της ουσίας και με βάση την οδηγία να πάρετε μια δίκαιη στάση, να είστε πιο ελαστικοί και πιο δραστήριοι. Άγκατα, μας πάτε ξεκάθαρα τι περιθώρια χειρισμών έχουμε. Οπότε ας την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, ώστε οι πολίτες της Ρουμανίας να έχουν την αίσθηση ότι το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στο πλευρό τους και ότι παίρνουμε σοβαρά το πρόβλημά τους. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να δώσω εγγυήσει ότι η ρουμανική κυβέρνηση θα το δει όλο αυτό με θετική ματιά Αν προκύψει κάποιο είδου κρίση, θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά, αλλά σε πρώτη φάση προτείνω να την αφήσουμε ανοιχτή, να στείλουμε την επιστολή, να ασκήσουμε πίεση στην ρουμανική κυβέρνηση και να δούμε τι θα συμβεί από εκεί και στο εξή. Ποια είναι η άποψή σας, συνάδελφοι. Είναι δεκτό αυτό. Μου φαίνεται πως ναι. Λοιπόν, σας ζητάω συγγνώμη αν το δούμε αυστηρά, το θέμα θα πρέπει να την κλείσουμε την αναφορά, όμως επειδή μπλέκεται και ψυχολογικός παράγοντας, ας το κάνουμε αλλιώ. Και άλλη ακόμα μία αναφορά που έχουμε είναι στο σημείο 30 της Μεσής Διάταξης τη Μόνικα Λαγκονίσκα ε, από τον ορισμό διαβίου εκπαίδευσης για την απειλή που δέχονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Πολωνία. Είναι παρούσα η αναφέρουσα και θα της δώσω τον λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνει να παρουσιάσω τον αφορά μου. Σας ευχαριστώ επίσης για την υποστήριξή σας πιο αργά παρακαλούμε, δεν μεταφράζεται η μιλήτρια τόσο γρήγορα που μιλάει. Dziękuję Σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση, λέει η αναφέρουσα. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την αναφορά, μεγάλη μας χαρά είμαστε εδώ από το Σεπτέμβριο του 2017 έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και η κατάσταση όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, όσον αφορά ε, ΜΚΟ, όσον αφορά άλλους φορείς που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία της ε, σημερινής κυβέρνησης, ε, η κατάσταση λέγω, έχει, έχει, έχει επιδεινωθεί γιατί δεν μιλούμε καν για την αυτονομία δράσης. Μιλούμε για τις δυσκολίες που έχουμε για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής γιατί συνεχώς νομοθετεί η κυβέρνηση χωρίς να τη νοιάζει τι σκέφτεται για αυτά που κάνει, τι σκέφτεται ο κόσμος. Το κοινοβούλιο της χώρας κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα. Πολύ λίγοι φορείς παίρνουν ε, κρατική υποστήριξη. Πώς να τους ανταγωνιστείς. Και όσον αφορά την κυβέρνηση, έχουμε διαμαρτυρίες που όμως κατευθύνονται από έξω ε, έχουμε κόσμο να διώκεται και να συλλαμβάνεται είχαμε 625 δικαστικές έρευνες και 333 αποφάσεις καταδικαστικές τα τελευταία μισή χρόνο είχαμε ένα σωρό διώξεις κατά διαδηλωτών Κάθε μήνα έχουμε 100 καινούργιες υποθέσεις τέτοιες. Όλα αυτά για διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση ελευθερίας του τύπου του 2017 πρόκειψε ότι η Πολωνία είναι η πρωταθλήτρια χειρότερα από το Μπουρούντι, τον Μπελίζε και την Τουρκία. Πολύ λίγες χώρες τα πήγαν χειρότερα από την Πολωνία. Και έχουμε και άλλα στατιστικά κατατείνουν στο ότι δεν πρόκειται περί δημοκρατικής χώρας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καταστήλει, να καθυποτάξει τους πολίτες και θέλει να καθιδρύσει αστυνομικό κράτος Έχουμε το νόμο του 2016 όσον αφορά την εισαγγελία και όσον αφορά ε, έναν καινούργιο αντιτρομοκρατικό νομό που έκανε τα πράγματα χειρότερα. Η εισαγγελία με αυτό το νέο νόμο έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Και όσον αφορά την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, πλέον δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την συλλογή δεδομένων όσον από πλευρά Ιντερνετ και τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει περιορισμό ε, και περιστολή του δικαιώματο ε, της διαδήλωση επίση. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση γιατί η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτού που δεν συμφωνούν ιδεολογικά μαζί τη. Έχει απελπιστεί ο κόσμος. Τον Οκτώβριο του 17 ο Πιότερ Τσέσνη ε, αυτοπυρπολήθηκε στο κέντρο της Λισαβόνας. Δέκα μέρες μετά εξέπνευσε. Θεωρούμε ότι έτσι δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει υγιής πολιτικός βίος. Είναι ξεκάθαρο ότι πια δεν χρειαζόμαστε εκθέσεις, χρειαζόμαστε ανάληψη δράσης. Έχουμε το άρθρο 7 που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί κατά Πολωνίας και Ουγγαρίας. Πάντως το βασικό είναι η κρίση χρηματοδότησης. πώς θα μπορέσουν οι μικρότερες οργανώσεις να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως Ευρωπαία, ως πολίτες της Ένωσης. Παρακαλώ, ακούστε μας. Και τελειώνουμε ένα ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως ε, ΜΚΟ για να σώσουμε την κοινωνία των πολιτών, να σώσουμε τη χώρα από ένα τέτοιο κόμμα σαν αυτό που κυβερνά. Μπορεί να κάνει τίποτα η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσει και εμάς και μη και όσοι άλλες χώρες για να στηρίξουν το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα. Το 2018 πού μπορούμε να στραφούμε για να προστατεύσουμε κράτος δικαίου και δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Κυρία, η κυρία Λίντα Ράμπο είναι εδώ και εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την αναφέρουσα για το γεγονός ότι μοιράστηκε μαζί μας τις ανησυχίες της αυτής. Θέλουμε να σας επισημάνουμε τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνουμε και στην ε, απάντησή μας στην αναφέρουσα. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί το βασικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Αποτελεί προαπαιτούμενο για μια υγιή δημοκρατία και τη χρηστή χάραξη πολιτικής. Η Κομισιόν γνωρίζει και ανησυχεί σοβαρά σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε μια σειρά από κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και δεσμεύεται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι, μας, ε, από το χέρι της για να προστατεύσει αυτόν τον χώρο. Η συζήτηση για την προστασία, την πρόθεση και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και τις ευθύνες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα θα ε, προωθηθεί και από την Κομισιόν στο ετήσιο κολόκιουμ που θα διοργανώσει η Κομισιόν για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και που θα διοργανωθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Πράγματι, ο χώρος της κοινωνία των πολιτών πρέπει να προστατεύεται και να προωθείται και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να το κάνουν αυτό. Καμία νομική πράξη δεν μπορεί να περιορίσει το χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εμποδίζοντα τι να εκτελούν θεμητά καθήκοντά τους ή θέτοντας ε, απαγορευτικά όρια στο έργο τους. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη σχετικά με τον ε, ρόλο και τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ως θεματοφύλακας της συνθήκης αναλύει τις νομικές πράξεις που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο υπό το φως των απαιτήσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βεβαίως δεν διστάζουμε να αναλάβουμε και δράση όταν θεσπίζεται νομοθεσία η οποία μπορεί να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που απορρέουν από το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο όπως συνέβη πρόσφατα στην Ουγγαρία για τις οργανώσεις και τις κοινωνίες των πολιτών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Βεβαίως, το μόνο που μπορεί να κάνει η Κομισιόν ε, ε, ε εντάσσεται, ε, αυτά που μπορεί να κάνει η Κομισιόν περιγράφονται και περιορίζονται από τις αρμοδιότητες της όπως αυτές κατοχυρώνονται στις συνθήκες. Δεν έχει γενική αρμοδιότητα η Κομισιόν να παρέμβει στα ίδια τα κράτη-μέλη, στο εσωτερικό των κρατών μελών, όταν υπάρχουν ε, καταγγελίε για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκτό εάν εμπλέκεται κάποια ευρωπαϊκή νομική πράξη. Και εδώ ε, μιλάμε για το, το δικαίωμα του συνέρχεσαι, της ε, ελεύθερης έκφρασης, του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή όταν αυτά τα θέματα πλήττονται, όταν υπάρχουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς, τότε μπορεί να αναλάβει δράση η Κομισιόν. Τώρα, συγκεκριμένα για την κατάσταση που περιγράφει η αναφορά, η Κομισιόν σημειώνει με ανησυχία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών στην Πολωνία. Ωστόσο, θέλει να τονίσει ότι όσον αφορά την πρόσβαση και την διασπορά, την, διανομή, την κατανομή ε, δημόσιων κονδυλίων σε οργανώσει κοινωνία των πολιτών, αυτό είναι ένα θέμα που εναπόκειται και εντάσσεται στις εθνικές αρμοδιότητες. Όσον αφορά την πολωνική πράξη για την ε, ίδρυση ε, ε, ενός πολωνικού ιδρύματος ελευθερίας που αναφέρεται ρητός στην αναφορά, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι συζητήσαμε το θέμα αυτό το Φεβρουάριο του 2018 με τις πολιτικές, πολωνικές αρχές για να λάβουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το ρόλο που προβλέπεται να έχει αυτός ο νέος οργανισμός, ιδίως όσον αφορά την ε, αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι πολιτικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι το Ινστιτούτο αυτό δεν συνδέεται με την κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων και μας ενημέρωσαν ότι θα εγκριθεί εκτελεστική πράξη η οποία θα καθορίζει το ρόλο ε, του συγκεκριμένου Ινστιτούτου και εκεί όταν θα εγκριθεί ε, αυτή η νομική πράξη θα ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Επίσης σημειώνουμε την κοινή γνωμοδότηση που εξέδωσαν ο ΣΑ και η Επιτροπή της Βενετίας και εκφράζει την ελπίδα της οι πολωνικές αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από διάφορες πλευρές σχετικά με την νομική αυτή πράξη. Ελπίζω ε, αυτά να δρουν διευκρινιστικά, να φώτισα το θέμα από πλευράς Κομισιόν και βεβαίω είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, λαμβάνω το λόγο από πλευράς του συνάδελφου Βαλέσσα. Θα σας πω και στο την προσωπική μου άποψη. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τη δημοκρατία και οι κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο ε, εφαρμόζουν τις διεθνείς αρχές για την προστασία των ΜΚΟ. Έχουμε διάφορες ε, διεθνείς συμφωνίες. Τις έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη υπό την αιγύδα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλοι δικαιούνται να συγκροτήσουν τέτοιες οργανώσεις για ειρηνική διαμαρτυρία, για έκφραση απόψεων. Κατόπιν της κατάργησης της εξαρτησίας δικαιοσύνης και κατόπιν της ε, καθυπόταξης των, των ε, ΜΜΕ στράφηκε η κυβέρνηση Πολωνίας κατά της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό για το κράτος δικαίου. Πέρσι η κυβέρνηση της χώρας έφτιαξε μια οργάνωση ούτως ώστε να κόψει κάθε χρηματοδότηση προς τις ΜΚΟ. Το Ίδρυμα Ζητημικής Ελευθερίας ε, τώρα αποφασίζει ποιες ΜΚΟ πρόκειται να τύχουν κρατικής επιχορήγησης. Η κυβέρνηση του νόμου και της δικαιοσύνης τώρα έτσι καθορίζει ποιος θα χρηματοδοτηθεί. Με αυτόν τον έλεγχο στον προτιμοδοτή των ΜΚΟ, το, η κυβέρνηση παρεμποδίζει το έργο τους. Τουλάχιστον για τις ΜΚΟ με τις οποίες διαφωνεί. Και έχουμε ένα σωρό ανησυχητικά τέτοια παραδείγματα. Αυτό το Ίδρυμα Εθνικής Ελευθερίας έκοψε χρηματοδότηση προς ΜΚΟ, τον οποίο το έργο δεν αρέσει στην ε, κυβέρνηση. Για παράδειγμα, δημιουργιωμάτων δημιουργιωμάτων των γυναικών, των μειονοτήτων. νομική παιδεία, παιδεία στους ε, κοινωνικούς πολιτικούς θεσμούς, όλα αυτά τα θεωρούν απειλή. Θέλουν να ισοπεδώσουν τις ΜΚΟ, θέλουν να ελέγξουν ε, τα πάντα. Η κυβέρνηση διαλέγει τους ευνοουμένους της για να υποστήριξει. Όμως για μια ανεξάρτητη χώρα είναι απαραίτητο όλες οι ΜΚΟ, όχι μόνο οι βελικές στην κυβέρνηση. Χρειάζεται μια πλουραλιστική κοινωνία. Ανεξάρτητη. Αυτή είναι η προϋπόθεση μιας ε, δημοκρατίας που λειτουργεί με υγιή τρόπο. Οποιαδήποτε δράση που περιστέλει την ελευθερία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανωσιών της. Κάθε απόπειρα ελέγχου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα σοβαρά. Γι' αυτό παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί το τι κάνει η πολωνική κυβέρνηση. Ό,τι, ό,τι κατατείνει στον έλεγχο των ΜΚΟ ε, προέρχεται από μια οπτική γωνία για έναν μονοδιάστατο κόσμο. ουσιαστικά αποκλείει τον κόσμο από τη συμμετοχή στην προβληματική για θέματα που άμεσα τον αφορούν. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Η κοινωτική χρηματοδότηση πρόκειται να πάει σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Πρόκειται για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μία εφημερίδα ιδεολογικά κοντά στην κυβέρνηση έχει στο δικαίωμα του Συμβούλιο έναν ευρωβουλευτή. Έτσι μπόρεσε αυτή η εφημερίδα να αποσπάσει αυτή τη χρηματοδότηση. Να, παράδειγμα για το πώς χρησιμοποιούνται τα κοινωτικά κονδύλια στην Πολωνία. Έχει έρθει σε επαφή η κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Νορβηγίας. Ε, γιατί η Νορβηγία διαφώνησε με τον τρόπο που τα δικά της χρήματα θα τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση της χώρας. Πρόεδρος. Θα θέλω να πάρουμε το λόγο Ποιος θέλει άλλος να πάρει το λόγο μάλλον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είναι μια μη πολωνική φωνή που θα υποστηρίξει αυτό που είπε Πετέρα σε αυτή την επιτροπή και είναι πολύ βασικό στις αξίες και στη δημοκρατία μας να διασφαλίσουμε ότι στις χώρες μας έχουμε πλουραλιστικά πλουραλιστική και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών. Το κίνημα περιορισμού της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι πολύ ανασχετικό όχι μόνο στην Πολωνία. Η Πολωνία όμως είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλες χώρες. στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και το λέω αυτό σαν ευρωβουλευτής που ενδέχεται να φύγω από αυτό το κλαμπ πριν τις επόμενες εκλογές το πρόγραμμα, το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα με τον διάλογο που έχουμε για την Ουγγαρία, με αυτά που συμβαίνουν στην Πολωνία, ε, και αυτό που στέλνω στην τελευταία ολομέλεια. Αν δεν έχουμε τις εξουσίες τις απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ε, την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τότε θεωρώ ότι σε αυτό το διάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα η Επιτροπή θα έχει συζητήσει τον επόμενο μήνα, αλλά θα πρέπει να γίνει συζήτηση για την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας απογοητεύει είναι ότι ναι, κάνουμε το διάλογο για την Πολωνία. Συζητήσαμε γι' αυτό στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Είχαμε διάφορες εκθέσεις για την κατάσταση και παρόλα αυτά πάντα αυτό που μας κρατάει πίσω είναι η έλλειψη εργαλείων, μέσων για να διασφαλίσουμε ότι οι θεμελιώδεις αρχές ε, προστατεύονται. Χρειάζεται να αναλογιστούμε ε, την κατάσταση, να δούμε πώς θα πρέπει να είναι αυτή η εργαλειοθήκη η ισχύς του ευρωπαϊκού εγχειρήματο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και να υπάρχει σεβασμός ε, ε, στο ρόλο που παίζουν ε, οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών στο εθνικό επίπεδο. Να δείτε και το επόμενο θέμα που έχουμε στη Μεσή Διάταξη για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τον ρόλο που έχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει σε αυτό το θέμα. Αν δεν ανθίσει η κοινωνία των πολιτών, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει συνοχή σε αυτά που λέω. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι ότι δεν θέλω μία τέτοια σημαντική αναφορά να έχει απαντήσει μόνο από λονούς πολιτικούς. Φυσικά είναι πολύ μεγάλη ανησυχία ε, για τις πολωνικές ε, μη κυβερνικές οργανώσεις και τις μυριζόμαστε πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο, άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, από κοινού την Επιτροπή, για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, Επιτρέψτε μου τώρα να αλλάξω λίγο το καπετελάκι μου και να πάψω για ένα λεπτό να είμαι προεδρεύων της συνεδρίασης. Θέλω λοιπόν εκ μέρους του ΕΛΚ να πω τα εξής. Λυπούμαστε βαθύτατα για το γεγονός ότι καλούμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε της άποψης ότι οι οργανώσει κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι ελεύθερες κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Βρισκόμαστε λοιπόν με το μέρος της αναφέρουσας, υποστηρίζουμε και εμείς την πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Εκφράζουμε δε και την υποστήριξή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις προσπάθειές της να βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλει ενδεχομένως η αναφέρουσα τον λόγο για να ξανατοποθετηθεί. Ε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που εκφράσατε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να είχε συζητηθεί το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή σας. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Διότι αυτό που είπε και μία από τις προλαλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην, Στην Πολωνία δεν έχουμε πια εργαλεία για να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχουν ούτε ευρωπαϊκά εργαλεία, μα πού θα τα βρούμε εν τέλει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η προηγούμενη κυβέρνηση πίστευε στην Ευρώπη. Η τωρινή δεν πιστεύει στην Ευρώπη. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ως πολίτες της Πολωνίας. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την, για την υποστήριξή σας και θέλω πραγματικά να σας ε, καλέσω να εξασφαλίσετε και εσείς την ισότιμη μεταχείριση και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Γιατί μόνο τότε και μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πραγματική, μια γνήσια δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί από την πλευρά μας η διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όποτε υπάρχουν, υπάρξουν νέα, θα πρότεινα να επανέλθουμε στο ζήτημα. Συμφωνείτε κι εσείς? Ωραία. Επομένως, Όσοι έχετε παρακολουθήσει από, την από το πρωί τη συνεδρίασή μας, μπορεί να εκπλαγείτε γιατί δεν μας έμεινε καθόλου χρόνος για διάλειμμα. Ξεκινάμε κατευθείαν με το επόμενο θέμα. Καλό τον κύριο καθηγητή να έρθει και να καθίσει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 Uh, Συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητοί συμμετέχοντες, είναι μεγάλη μου χαρά που έχω τη δυνατότητα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση σχετικά με τα δικαιώματα των αναπήρων που ε, διοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε χρόνο λοιπόν ε, διοργανώνουμε ως Επιτροπή μια τέτοια ακρόαση. Είναι η τέταρτη φορά που θα ακούσουμε εμπειρογνώμονες και θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με, ε, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες τεχνικού χαρακτήρα πληροφορίες. Η ακρόαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και οι παρεμβάσεις των ομιλητών και των συμμετεχόντων θα καταγραφούν. Έχουμε διερμηνείς ε, και στην νοηματική γλώσσα. Και θέλω όσους τα χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν και τις ε, σχετικές συσκευές που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω επίσης να καλωσορίσω την κυρία Καμπεθόν, την συνάδελφό μου, η οποία και θα προεδρεύσει του πρώτου πάνελ ομιλητών καθώς και την κυρία Φαραγκούτ που θα προεδρεύσει του δεύτερου πάνελ. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Μάρκ Πρέστλε που είναι καθηγητής ε, πολιτικής για τα άτομα με ανεπηρίες και επιστημονικός διευθυντής του Ακαδημαϊκού Δικτύου ε, Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ατόμων με αναπηρία. Έχετε 15 λεπτά τον λόγο κύριε Πρέστλε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που μου απίφθηνε για να σας ενημερώσω και να συγχαρώ επίσης την Επιτροπή για την ετήσια αυτή εκδήλωσή της για ένα τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα σχετικά με τη σημασία που έχει το θέμα αυτό. Η παρουσίασή μου λοιπόν αφορά μια επικαιροποίηση της μελέτης που σας παρουσιάσαμε πριν από τέσσερα χρόνια και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την λήψη ε, υπόψη της διάστασης των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα του έργου της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο ε, της ε, Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Επιτροπή Αναφορών λοιπόν ανέθεσε σε εμά το 2015 να εκπονήσουμε μια μελέτη με την οποία να θα αναλύαμε ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Βεβαίως προβλήματα ε, των ατόμων με αναπηρίες είναι μια πολύ ευρία έννοια, αφορά την φτώχεια, την απασχόληση, την, ε, το δομημένο περιβάλλον, τις διακρίσεις, είναι πάρα πάρα πολύ ευρύ το θέμα βεβαίως. Εμείς λοιπόν επικεντρωθήκαμε σε εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται ε, με τις αναπηρίες και που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή κοιτάζουμε την ε, αναπηρία όχι μέσα από το πρίσμα της ατομικής υγείας αλλά μέσα από το πρίσμα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής αυτό. Όταν μιλάμε λοιπόν για αναφορές που σχετίζονται με, την, με τις αναπηρίες σε αυτόν τον τομέα και σε αυτή τη διάσταση ε, αναφέρομαστε. Επίσης κοιτάξαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την συμπερίληψη της διάστασης των ε, δικαιωμάτων των ε, ατόμων με αναπηρία σε όλο το έργο των θεσμικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και, δυστυχώς, ευτυχώς μπορώ να, σας ενημερώσω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και φυσικά σε αυτή τη θετική πρόοδο έχει συμβάλει και η Επιτροπή Αναφορών, η δική σας Επιτροπή. Στην αρχική μελέτη λοιπόν εξετάσαμε το πλαίσιο ε, της σύμβασης του ΟΗΕ για τα, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Και παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή σας λαμβάνει πολλές αναφορές, βεβαίως, σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τις, αναφορ, με αναπηρίες, έχει και συγκεκριμένες, αν θέλετε, νομικές ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είναι συμβαλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ταυτόχρονα όλα τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης αυτής. Είναι διεθνής η σύμβαση αυτή. Και μία από τις ε, ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή είναι η προστασία, η προώθηση και η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η Επιτροπή Αναφορών έχει συγκεκριμένη λοιπόν ε, ευθύνη μέσω της διαδικασίας των αναφορών ε, στην προστασία των, και την προώθηση, θα έλεγα εγώ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτά τα θέματα, ε, θα σας ε, παρουσιάσουμε κάποια παραδείγματα και θα διατρέξω και εντάχει ε, κάποιες συστάσεις μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα αρκετά περίπλοκο ε, περιβάλλον από άποψη πολιτικής. Έχουμε το διεθνές πλαίσιο, τη σύμβαση, το διεθνές δίκαιο, έχουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, έχουμε εθνικές στρατηγικές στον ίδιο τομέα και έχουμε και τις τοπικές ε, πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι η ε, ε, τα άτομα με αναπηρίες ε, είναι μια πολύ μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα. 25% του εκλογικού σώματος στην Ευρώπη ε, αναφέρει ότι έχει κάποια αναπηρία Επομένως είναι ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ ισχυρό αν θέλετε εκλογικό σήμα. Στην αρχική μελέτη παρατηρήσαμε ότι πολλές από τις απαντήσεις που δίνει η Επιτροπή σας ε, δεν έχουν δικαστικό χαρακτήρα αν θέλετε, δεν είναι εκτελεστές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Επιτροπή σας και γι' αυτό η σύσταση προς την Επιτροπή σας ήταν να συνεχίζετε να ασκείτε πίεση στις εθνικές αρχές, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή με τους ήπιου και λιγότερο ήπιου, αν θέλετε, τρόπου που έχετε στην διάθεσή σα. Οι αναπηρίες λοιπόν εξακολουθούν ένα πολύ πιεστικό ζήτημα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που, απασχολούν την, που απασχολεί την Επιτροπή σας. Πολλές αναφορές αφορούν την, τις, τα άτομα με αναπηρίες, η αναλογία λοιπόν των αναφορών που αφορούν τις ε, αναπηρίες δεν έχει αλλάξει, αν και υπάρχει μια μικρή διακύμανση, αλλά είναι, είναι, είναι σχετικά λίγες. Όμως οι αναφορές αυτές που αφορούν τα άτομα με αναπηρίε έχουν ιδιαίτερη νομική βαρύτητα, γιατί συνδέονται με δικαιώματα που απορρέουν από διεθνεί συμβάσει. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτέ τι αναφορέ να τι λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Οι πλέον ε, συνήθεις ε, αναφορές αφορούν ζητήματα προσβασιμότητας, κοινωνικής προστασίας, δικαιωμάτων στην εργασία, αλλά και το δικαίωμα να μπορεί κανείς να ζει ανεξάρτητα στην τοπική κοινωνία του και να απολαμβάνει και κοινοτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά την ε, προσβασιμότητα, εδώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται οι περισσότερες αναφορές που έχετε λάβει. Οι που έχουν εκφράσει πολίτες για μην, ε, την αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση σε δημόσια μέσα συγκοινωνίας, σε δημόσιες εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια. Υπάρχουν επίσης μια σειρά από ε, μια σειρά από όπου μπορεί να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, μιλώ για παράδειγμα για τη δέσμη μέτρων για τις μεταφορές. Και εδώ έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος. Ασκήσατε λοιπόν πίεση ως Επιτροπή με τις συστάσεις σας για να σημειωθεί αυτή η πρόοδος και να εγκριθεί η ευρωπαϊκή πράξη για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο του τριμερούς διαλόγου. Έχετε αποστείλει και συγκεκριμένες συστάσεις και γνωρίζω ότι το Συμβούλιο ενέκρινε θέση που με κάποιο τρόπο αποδυναμώνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό ε, ίσως σημαίνει ότι οι υποσχέσεις που έχετε δώσει σε διάφορους αναφέροντες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εκπληρωθούν πλήρως παρόλα αυτά όμως ε, ε, πρόκειται για πρόοδο. Στην απασχόληση δέχονται διακριτική μεταχείριση τα άτομα με αναπηρίε. Φαίνεται ότι ε, και ο κοινωνικός πυλώνα όμως έχει ε, επιφέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Ε, κινητοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν κάποια επιχειρήματα μέσω της σύστασης αυτού του κοινωνικού πυλώνα βελτιώθηκαν τα πράγματα και πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διάφορου τομεί πολιτική και νομίζω ότι και η Κομισιόν έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να συμπεριλαμβάνεται αυτή η διάσταση στι πολιτικέ τη για την απασχόληση αλλά και άλλου τομεί πολιτική. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικό η Κομισιόν να συνεχίσει να ε, ε, επιστήνει την προσοχή των αρμοδίων σε παραβιάσει μέσω από τα εργαλεία που έχει γίνει στα χέρια τη, ε, το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό εξάμεινο κτλ. κτλ. Και τέλος, κοινωνική προστασία, επίπεδο, βιωτικό επίπεδο. Βλέπουμε αναφορές που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία, με τα συστήματα επιδομάτων, ε, αναπηρικών συντάξεων κτλ. Γνωρίζουμε από την Επιτροπή του ΟΗΕ ότι, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί, θεσπιστεί πολλές πολιτικές λιτότητας που περιόρισαν τα επιδόματα, ε, που έρχονται, πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση ακόμη και με συγκεκριμένα άρθρα της σύμβασης, όπως είναι το άρθρο 26. Ε, το Ηνωμένο ε, Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει κατηγορηθεί ως ε, ότι προβαίνει σε συστηματική παραβίαση της σύμβαση των ατόμων για τα δικαιώματα των ατόμων με, με αναπηρίες. Βεβαίως, υπάρχει κοινή, αρμοδιο, κοινή αρμοδιότητα, πολλά θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, άλλα θέματα εμπίπτουν, είναι κοινή αρμοδιότητα κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση ε, και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδο. Ε, όσον αφορά την, ανεξάρτητη, τη δυνατότητα να ζήσει κανεί ανεξάρτητα στην τοπική του κοινωνία, έχουν υπάρξει κάποιε πολύ σημαντικέ αλλαγέ ε, ε, τα τελευταία χρόνια σε ορισμένε χώρε όπω είναι η Φιλανδία. Ε, και νομίζω ότι και η δική σας στάση ήταν πολύ θετική στην, στις επαφές σας με τις φιλανδικές αρχές, βλέποντας από τις ε, απαντήσεις που σας απέστειλαν οι φιλανδικές αρχές, ε, πράγματι έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη ε, τους τις συστάσεις της Επιτροπής σας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα αυτό το ζήτημα ε, της ε, αποϊδρυματοποίησης, μέσω, των μέσω των πολιτικών συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έργο που έκανε και ο Φρά στο άρθρο 19 και θα σας το παρουσιάσει και σε λίγη ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος, μιλάμε για τη συμμετοχή στην πολιτική κοινωνική δημόσια ζωή. Δεν υπήρξαν πολλές αναφορές για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω ότι επίκυνται οι ευρωεκλογέ το 2019 και εκεί σε συνεργασία με τον ΦΡΑ καταφέραμε να προσδιορίσουμε συστηματικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκλογικών δικαιωμάτων ε, στις τελευταίες εκλογές ατόμων με αναπηρίε πάντοτε. Και εδώ νομίζω ότι έχετε το ρόλο να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει ε, προκειμένου να απευθυνθούν αντίστοιχε παραβιάσεις τη εκλογική νομοθεσία στις εκλογέ του 2019. Ήδη υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται για το τι θα κάνουν σε περίπτωση που τους, που τους ε, ε, αρνηθούν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία λόγω αναπηρίας στις εκλογές του 2019. Υπήρξαν πάντως σε κάθε περίπτωση αρκετές αλλαγές. Ο Μακρόν στη Γαλλία ανακοίνωσε ότι στις επικείμενες εκλογές θα έχουν το δικαίωμα ψήφου όλοι οι Γάλλοι πολίτες Μόνο όμω μικρό ποσοστό των κρατών μελών μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι ε, εξασφαλίζει πραγματικά το δικαίωμα, το εκλογικό δικαίωμα σε όλους τους ε, πολίτες τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να συμπεριληφθεί αυτή η διάσταση της αναπηρίας σε όλο το έργο του Κοινοβουλίου, όχι μόνο στη δική σας Επιτροπή, στην Επιτροπή Αναφορών. Όπως ε, εξηγούμε και στο επεξηγηματικό σημείωμα, βεβαίως αναγνωρίζουμε τη δραστήρια ε, συμμετοχή σας ε, σε διάφορα φόρα, σε διάφορα μέτωπα και μετερίζια που συζητείτε αυτό το θέμα Ξέρω ότι πολλά μέλη τη Επιτροπή Αναφορών συμμετέχουν και σε άλλε επιτροπέ και εκεί θέτουν το ζήτημα. Δεν έχουμε ακόμη ε, καταφέρει να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψη τη διάσταση τη αναπηρία όπω έχουμε καταφέρει να, να, την εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψη τη διάσταση του φύλου, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά σημειώνεται πρόοδο και αυτό το χρεώνεται, το πιστώνεται μάλλον και η δική σα Επιτροπή. Για παράδειγμα, μόνο η Επιτροπή Γεωργία είναι. Ε, ε, που δεν έχει ακόμα ασχοληθεί με, το ζήτημα των, ατόμων, των δικαιωμάτων των ατόμων με ανεπίρρε. Και αυτό είναι πραγματικά βήμα προ σωστή κατεύθυνση. Είναι πρόοδο. Το να λαμβάνονται υπόψη, να υπόψη τα άτομα με αναπηρίες σε όλε τι πολιτικέ. Όταν το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τις συστάσεις του ΟΗΕ αυτό αποτέλεσε μια πραγματικό κίνητρο ε, διακομματικά, διακοινοβουλευτικά. Υπήρχαν πολλές επιτροπές που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Λάβαμε ε, διάφορες προτάσεις, συστάσεις, καταλήξαμε. Χρειαζόμαστε άλλο ένα τέτοιο κίνητρο, αν θέλετε, άλλο ένα τέτοιο ερέθισμα για να ξαναξεκινήσει και να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη όθεση. Η προφανή όθηση θα δοθεί βεβαίω από την ολοκλήρωση και την οριστικοποίηση τη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Επίσης υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καθώς ε, πρόκειται να κυρώσει και το προοριτικό πρωτόκολλο που δίνει το δικαίωμα στα, στους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει, είναι μια κίνηση η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη δική σας Επιτροπή. Είναι μια ευκαιρία για να ενισχυθεί το πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της προστασίας, της παρακολούθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, να δοθεί ένας πιο συστηματικός και συνεπής χαρακτήρας στο πλαίσιο αυτό. Η επόμενη έκθεση ε, προόδου ε, θα εκδοθεί σύντομα και θα κοινοποιηθεί στον ΟΗΕ. Πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει μια επικαιροποίηση, μια ανανέωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία μετά το 2020. Μέσω του προϋπολογισμού λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλές ευκαιρίες για να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να σημειωθεί πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς πολιτικής ε, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν τα άτομα με αναπηρίες και τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 10 λεπτά για συζήτηση, αν έχετε ερωτήσει ή σχόλια να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάρκ για το θέμα της αναπηρίας και την προοπτική που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και ως το ως πώς θα προχωρήσει σε συστάσεις και δράσεις στο μέλλον. Αυτή την εβδομάδα μια από τις βασικές ειδήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια έκθεση από την Επιτροπή Ποιότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και είχαμε ε, τον εξής τίτλο ότι είναι στους πέντε ανθρώπους ε, στο Ηνωμένο Βασιλείο με αναπηρία ε, δέχονται παραβίαση δικαιωμάτων. Είναι πολύ άδικο αν επιβάλλονται μέτρα λιτότητας και το πώς έχουν αλλάξει τα συστήματα, τα επιδόματα με τέτοιο τρόπο ώστε να τιμωρούν ουσιαστικά νοικοκυριά και οικογένειες όπου ένα συνήλικας ή ένα παιδί ε, έχουν κάποια αναπηρία. Με εντυπωσίασε η ενα παιδι εχουν καποια αναπηρια διαφάνεια για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σχετικά με τις ιδέες που εκφράσατε για τις ευρωεκλογέ, για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Θεωρώ ότι το να αντιμετωπίσουμε ε, το, μακ, το μακροοικονομικό θεματολόγιο είναι πολύ θεμελιώδες, ώστε να μπορέσουμε να ε, βγάλουμε τους ανθρώπους με αναπηρία από τη φτώχεια, στο να εφαρμόσουμε δίκαιες πολιτικές και να καθιερώσουμε ένα πιο δίκαιο πλαίσιο όχι για να υπονομεύσουμε προσπάθειες ή δημιουργία μια σωστή νομοθετικής πράξης και σωστές δομές ώστε να μπορούν τα άτομα να συμμετέχουν Α, αλλά αυτό θα αποβεί ενάντια στα άτομα εμπειρία, αν συνεχίσουν να τιμωρούνται δυσανάλογα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό, αυτό ήθελα να τονίσω εξ αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια από αυτού. Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη. Τις τελευταίες τρεις μέρες ε, μελετούσα δεδομένα της Eurostat για τη στάση των τελευταίων δεκα ετών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την φτώχεια στα άτομα με αναπηρία όσον αφορά τους στόχους ε, για τη βιωσιμότητα είναι πολύ... Ε, υπάρχει ο κίνδυνος ε, να μείνουν πίσω τα άτομα με όταν ανακάμπτουμε οικονομικά και βλέπουμε αυτό το χάσμα, αυτή την ψαλίδα να διευρύνεται καθώς η κοινωνία ουσιαστικά επωφελείται από την βελτίωση της κατάστασης και κάποιες ε, ομάδες ατόμων να μένουν πίσω Μεγάλο ο κίνδυνος κατά τη διάρκεια της περίοδου λιτότητας, αλλά τώρα προκύπτουν και νέα, ε, νέοι κίνδυνοι ε, με την ανάκαμψη, ώστε ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα. Κύριε Κουνέδο Κύριε Κούρεβα, συγγνώμη. Ήθελα να, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κατηγητά. Εσείς βλέπετε πώς εξελίγουν τα ζητήματα της αναπηρίας. Οι περισσότερες χώρες έχουν περάσει ρυθμίσεις στην νομοθεσία τους. Αλλά δεν τηρείται καμία νομοθεσία και από εδώ περνάμε διάφορες ρυθμίσεις. Αλλά όλα αυτά δεν γίνεται πράξη. Να πάρουμε ε, Βρυξέλλες. Ένα πολύ απλό παράδειγμα και το βλέπουμε όλοι που δεν είναι καθόλου προσβάσιμο. Και είναι μια πόλη στην οποία πέφτουν πάρα πολλά λεφτά και δεν γίνεται καμία αλλαγή. Και εδώ είναι συγκεντρωμένοι όλε οι οργανώσει και ευρωπαϊκέ και παγκοσμίω και δεν υπάρχει καμία προσβασιμότητα. Και γύρω γύρω στο κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσει και να κινείσαι. Εσείς πώς βλέπετε, μπορείτε να προτείνετε κάτι. Okay. Maybe. Wilkins. Θα μπορούσατε να απαντήσετε στην κυρία... David Wilkins, να απαντήσετε στην κυρία Κούνεβα. Okay. Um, I would just... Λοιπόν, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο βασικός ομιλητής και η προελή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Βασιλείο και σε άλλες χώρες είναι ότι όταν βελούνται η οικονομική κατάσταση μένουν πίσω τα άτομα με αναπηρία και ένα παράδειγμα είναι ότι προσπαθώ να βρω δουλειά σε όλη μου τη χώρα χαίρομαι όμως που είμαι εδώ γιατί τώρα δουλεύω σε έναν εκπληκτικό οργανισμό Παρ' όλα αυτά όμως με απογοητεύει το γεγονός ότι δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στις Βρυξέλλες χρειάστηκε να φέρω έναν εκπαιδευτή που θα με βοηθήσει ώστε να μπορέσω να έχω πρόσβαση γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ προοδευτικό όταν πάντα μου λένε ότι το Ευρωκοινοβούλιο ε, θέλει να, να συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Θεωρώ ότι αυτή η Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την κατάσταση θα συμβεί όμως αυτό, δεν υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα ε, με τον ίδιο τον οργανισμό που προσπαθεί να το καταστήσει δυνατό. Bueno, Πρόεδρος, έχω δύο παρατηρήσεις. Μετά θα λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα πρώτα. Άκουσα τι ελέγχθη προηγουμένως όσον αφορά τον λόγο των ε, ε, αναφορών. Είναι σημαντικός ρόλος, πρέπει να τον αναβαθμίσουμε, να βοηθήσουμε τους αναπήρους και θα πρέπει για την απασχολησιμότητα, την προσβασιμότητα, τα γενικά θέματα να μπορεί κανείς να απευθύνεται σε εμάς. Ε, βέβαια και δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο προσβασιμότητα εδώ στο κτίριο. Να δούμε πώς και για άλλα θέματα αναφορές θα έρχονται. Γιατί δεν είναι και λίγες. Και θα πρέπει κάποιοι να μπορούν να έρθουν εδώ να πούν το πρόβλημά τους. Δεν έχουμε αναφορές για εκείνους από τους αναπήρους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Και εδώ μπορέσαμε να συζητήσουμε τι γίνεται με τους ανηλίκους. Πώς και αυτοί θα ακουστούν εδώ. Επίσης, να δούμε τι γίνεται επομένω και με τους ανηλίκους με αναπηρία. Πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμα και νομίζω βελτιώσαμε σε αυτή τη θητεία για την πρόσβαση μέσω του ίντερνετ για αυτούς που έχουν προβλήματα στην όραση. Νομίζω ότι οι πόρτες είναι ορθάνοιχτες εδώ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για τους ανθρώπους με αναπηρία. Μια ερώτηση τώρα. Όσον αφορά αυτό το οποίο έλεγε το πρώτο slide. Έχουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το εθνικό πλαίσιο. Έχουμε διάφορα πλαίσια. και διαφορετικά δικαιώματα, διαφορετικό τρόπο άσκηση των δικαιωμάτων ανάλογα με το που βρίσκονται τα εν λόγω πρόσωπα. Γι' ε, αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε. Ακούστε ένα παράδειγμα. Μιλάμε τώρα για τον χάρτη των προσώπων με αναπηρία, δηλαδή για το πώς μπορούν να μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος να μην υπάρχουν δεσμενές διακρίσεις και να υπάρχει ευκαιρία μετακίνησης αυτών των προσώπων. Άρα θα πρέπει όμως να έχουμε κάποια ελάχιστα κριτήρια εναρμόνισης. Τι θεωρείται αναπηρία. Να λύσουν τα οικονομικά θέματα. Προς το παρόν δεν έχει πει ποτέ όχι το Συμβούλιο και αρκούνται στις δικαιολογίες, στις αιτιολογίες μάλλον της πολιτικής μας. Άρα θα πρέπει να αναγνωριστεί η πολιτική αυτή, να αναγνωριστεί το πώς θα διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση αναπηρίας από όλους τους Ευρωπαίους. Κριτήρια αναγνώρισης της αναπηρίας. Να υπάρχει μια κάρτα και κάποιος παντού να αναγνωρίζεται να τον βοηθά αυτή η κάρτα τον ανάπηρο όπου πηγαίνει. Έτσι θα σημειώσουμε πρόοδο. Υπάρχει αντίσταση, υπάρχουν πολλοί φραγμοί. Αλλά αυθεντική αναθεώρηση της ε, ε, νομοθεσίας γίνεται μόνο έτσι. Έτσι θα παρακάμψουμε τον κίνδυνο της δυσμενούς διάκρισης. Εναρμόνιση κριτηρίων. Αναγνώριση ομοιογενός σε όλες τις χώρες. Αλλά δεν έχουμε ακόμα το νέο ορισμό. Στηριζόμαστε στα όσα προβλέπει ο ΙΕ. Χρειάζεται να προωθήσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Ας βρούμε λοιπόν αυτά τα κριτήρια που να είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες. και να μην υπάρχει πρόβλημα αν μετακινείται κάποιος με αναπηρία από το ένα κράτος μέλος σε άλλο. Χρειάζεται να γίνει αυτό με τα ομοιόμορφα κριτήρια. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Bueno, pues le damos la palabra a la Comisión Europea que quería intervenir. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay, thank you. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις αυτές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και για τη συζήτηση που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να κάνουμε. Το γεγονός ότι συζητούμε τα θέματα αυτά μας βοηθά πολύ όσον αφορά την ενίσχυση της, των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αναπηρία. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά θέματα βεβαίως και θέλω να πω ότι το ε, τρέχον έργο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Και αυτή σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε περίοδο ε, αξιολόγησης, ε, ενδιάμεσης αν θέλετε, για να δούμε τι τελικά στέφθηκε με επιτυχία, τι πρέπει να διορθωθεί, τι πρέπει να ενισχυθεί. Όσον αφορά την κάρτα αναπηρίας, είναι ένα μέτρο που το αξιολογούμε και εμείς ε, έχουν ε, βεβαίως υπάρξει κάποια πιλωτικά προγράμματα επιτυχημένα σε κάποια κράτη-μέλη. Θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε και να βεβαιωθούμε τι πράγματι απέφερε θετικά αποτελέσματα και τι περαιτέρω μπορεί να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τη διασύνδεση της αξιολόγησης ε, με, την, με τις πολιτικές αναπηρίας, Είπε και η Πρόεδρος ότι αυτό το θέμα ε, ε, έγκυται ε, εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό που προσπαθούμε όμως να κάνουμε στην Κομισιόν είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν τα μέτρα τους με τρόπο που θα είναι θα συμμορφώνεται με την σύνδεση, με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Μέσα των χρηματοπτικών μας ε, προγραμμάτων λοιπόν υποστηρίζουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να υπάρξει μια σύγκληση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα που ενδέχεται να άπτονται της επικουρικότητας. Είναι ε, θετικό και θεμητό βεβαίως ε, να υποστηρίζει η Κομισιόν πολιτικές και σύγκληση των πολιτικών σύμφωνα και με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Αυτή είναι η στάση μας και στους τριμερείς διαλόγους. Διευκολύνουμε την εξέβρεση συμφωνίας έως το τέλος του 2018. Να πω και δύο λόγια για την πολιτική συμμετοχή που επίσης αναφέρθηκε από τους ομιλητές. Θέλω να σας παραπέμψω στις συστάσεις της Κομισιόν που έγινε ε, εν ώψη των επικείμενων εκλεγών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά πλέον υπάρχει ε, αναφορά στα άτομα με αναπηρίες ε, και στο έργο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τι πρέπει να συμβεί. Λάβαμε σοβαρά υπόψη μας τη διάσταση της αναπηρίας. Όλα αυτά, οι γνώσεις που έχουμε πλέον σήμερα ε, για τα άτομα με αναπηρίες δεν θα τα είχαμε αν δεν είχε γίνει στατιστική δουλειά από την Eurostat. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από τη δουλειά αυτή να επιβεβαιώσουμε τα κενά που υπάρχουν και που διατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, ταυτόχρονα όμως ε, αναγνωρίζουμε ε, και σημειώνουμε ότι το, τα κενά αυτά δεν, διευρυ, δεν ευτυχώς στη διάρκεια της κρίσης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει και θα συνεχίσουμε βέβαια να παρακολουθούμε την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της συμπερίληψης της διάστασης αναπηρίας. Εκεί υπάρχει ο πυλώνας, όπου δεν αναφέρονται απλώς ρητό στα άτομα με αναπηρίες, έχουμε λάβει υπόψη μας πλέον τα ζητήματα που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία στην στέγαση, στην απασχόληση, στο περιβάλλον και σε μια σειρά από άλλους τομείς πολιτικής. Η συμπερίληψη αυτή της διάστασης της αναπηρίας πρέπει να ε, πραγματοποιηθεί σε όλες τις πολιτικές που θα χαράσσονται σε εθνικό, ε, ευρωπαϊκό, περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, η πρόοδος της συμπερίληψης συνίσταται στο γεγονός ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπέγραψε αυτή τη συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το παράρτημα της απόφασης του Συμβουλίου περιλάμβανε 40 νομικές πράξεις που αποτύπωναν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σύμβαση αυτή. Στην μελέτη προόδου που εκπονήθηκε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, ε, που επικεντρώθηκε στο τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Πριν από δύο χρόνια δημοσιεύθηκε. Ε, καταφέραμε και εντοπίσαμε πλέον 130 νομικές πράξεις που λαμβάνουν υπόψη τις και περιλαμβάνουν ε, ρητός ε, διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να εξασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι διατάξεις που πλέον έχουν θεσπιστεί θα εφαρμοστούν και με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτά και σας ευχαριστώ για όλες τις προφορίες που είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να ακούσουμε από τις παρεμβάσεις των ομιλητών. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το πρώτο ε, πάνελ. Να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές γιατί έχουμε και μια καθυστέρηση 10 λεπτών ήδη σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Πρώτο πάνελ λοιπόν αφορά την, τις νομικές ικανότητες των ε, ατόμων με αναπηρία και το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι μεγάλη μου ευχαριστησή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται και να τονίσω πριν τι επόμενε ευρωεκλογέ κάποιε προκύκλει και πόδια που υπάρχουν για του ανθρώπου με αναπηρία στο πολιτικό και το δημόσιο βίο. να συμμετέχουν στι εκλογέ, να εκλέγονται και να εκλέγουν και επίση να παρακολουθούν ε, τις ε, ειδήσει. Είναι πολύ δύσκολο να ζει κανεί σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή είναι πολύ ευρύ και δεν θα μπω σε λεπτομέρειε ή στι ε, νομικέ υποχρεώσει, ε, υπό το άρθρο 29 ε, του, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ. Αυτό που θέλω να σα θυμίσω είναι ότι αυτό το άρθρο το 29 επιβάλλει και αρνητικές υποχρεώσεις όπως να μην θέτονται όρια και εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου, αλλά και θετικές υποχρεώσεις, όπως είναι το υποχρεώσει να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν να παρακαμφθούν τα εμπόδια τα οποία μπορεί να εμποδίσουν τα άτομα ανεπηρία να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Μια από τις βασικές προκλήσεις, και θα όσο πιστεύω γίνεται, δείχνει ε, τα απορίσματα αυτά μέσω δεδομένων που έχουν αληθεί από το ε, Δίκτυο ε, Εμπειρογνωμόνων για θέματα αναπηρίας. Το 2014, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εκδώσαμε μία έκθεση για με την κατάσταση για την πολιτική συμμετοχή και θα επαναλάβουμε αυτό το έργο ε, στις επόμενες, ε, για τις επόμενες ευρωεκλογές. Ένα από τα βασικά πορίσματα του έργου μας είναι ότι πρώτον ότι τα άτομα με αναπηρία ενδιαφέρονται στο να συμμετέχουν στον πολιτικό βίο και στην πολιτική. Κατά πόσο αυτό ε, αντικατοπτρίζεται στην εκλογή τους σε πολιτικές ομάδες είναι ένα άλλο θέμα. Επίσης, να σας πω ότι θα πρέπει να προσέξουμε για τον τρόπο και τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων. Υπάρχει από το δεδομένα από δύο ευρωπαϊκές υπηρεσίες που ε, δείχνουν μια πολύ θετική εικόνα της κατάστασης γιατί δεν περιλαμβάνονται στις μετρήσεις αυτές τα άτομα που έχουν αναπηρίες που δεν τους εμποδίζουν να συμμετέχουν σε μια μεγάλη έρευνα πως είναι άτομα που έχουν ε, ψυχοκοινωνικές ε, αναπηρίες, άτομα που βρίσκονται σε ιδρύματα. Τα βασικά ευρήματα, όπως βλέπετε, είναι ότι πρώτον τα άτομα με αναπηρία ενδιαφέρονται για την πολιτική Υπάρχουν ε, διαφοροποίησεις ανάλογα με τις πολιτικές παραδόσεις ε, στα κράτη-μέλη και το πιο σημαντικό υπάρχει έλλειψη ε, συγκριτικών και αξιόπιστων στοιχείων. Οι στατιστικές φαίνονται εδώ και βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη στη Σλοβακία και στην Ιρλανδία υπάρχει ένα κενό μεταξύ ατόμων με αναπηρία και αυτών χωρίς όσον αφορά το ενδιαφέρον για την πολιτική και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την ε, πραγματική συμμετοχή και υπάρχουν πάλι σημαντικά κενά για άτομα με αναπηρίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ε, ηλικιωμένου που έχουν ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές, στις εκλογές από ό,τι άτομα χωρίς αναπηρίες. Φαίνεται και πάλι ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα ότι τα άτομα με θέλουν να συμμετάσχουν, όμως υπάρχουν βασικά εμπόδια. Και ποια είναι αυτά τα εμπόδια. Στην διαφάνεια που βλέπετε, λοιπόν, βλέπετε κάποια από αυτά τα εμπόδια. Πρώτον, τα εμπόδια που αφορούν τη νομική τους ικανότητα, τα ε, νομικά και διοικητικά εμπόδια, οι περιορισμοί για άτομα με διανοητικές αναπηρίες και προβλήματα. Αυτός ο στενό δυσμός μεταξύ νομικής ικανότητας και του δικαίωματος ψήφου αφορά όχι μόνο το δικαίωμα ψήφου αλλά και το δικαίωμα να εκλεγεί κανείς. Δεύτερον, τα άτομα με αναπηρίες αν κοιτάξετε αριστερά, αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν την προσβασιμότητα. Η μητέρα μου τη ζητήθηκε να πάει στο δεύτερο όρφο για να ψηφίσει, ενώ βρισκόταν σε αναπηρικό μαξίδιο, κάτι που ήταν αδύνατον. Ε, δεν μπορούσε να α, ε, ψηφίσει στο ισόγειο και χρειάστηκε να την κουβαλήσει κάποιο αστυνομικό ε, στον πάνω όρφο, κάτι που προφανώς στείλει την αξιοπρέπειά της. Έτσι λοιπόν προβλήματα προσβασιμότητας υπάρχουν παντού και είναι πολύ κοινά. Υπάρχει και έλλειψη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μεταξύ βασικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών και στα πολιτικά κόμματα και στις δημόσιες αρχές και, τους, ε, και τα μέσα ενημέρωσης για το πώς μπορούν να καταστήσουν τα μηνύματα ε, τους πιο σαφή και τι διαδικασίε πιο προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Το, τρίτο, το τελευταίο πρόβλημα αφορά την ε, συμμετοχή. Θα σα θυμίσω την συζήτηση που προηγήθηκε για την, το σημαντικό ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τη για την ε, άσκηση και την επιβολή τη δημοκρατία, Τα άτομα με αναπηρία σε διαδικασίες λήψη αποφάσεων είναι πολύ σημαντικά και όταν μιλάμε για συμμετοχή κάνουμε ε, Μιλάμε για συμμετοχή των οργανώσεων που τις εκπροσωπούν ε, στην πολιτική διαδικασία, το να μπορούν ε, να εκλεγούν στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στα τοπικά κοινοβούλια είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα βασικό δικαίωμά τους. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ένα θέμα που προκύπτει ε, επανειλημμένος στην έρευνά μας που αφορά την έλλειψη συστηματικής συλλογής δεδομένων οι οργανώσεις ε, ατόμων με αναπηρία και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο ώστε να ε, αφυπνίσουν φορείς σε εθνικό επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία και για το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα ώστε να ε, μεταφέρουν τα μηνύματά τους. Όσον αφορά τις χώρες, κοιτάζοντας τα κράτη-μέλη και την νομοθεσία και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ρευστότητα γιατί η νομοθεσία αλλάζει αλλά γενικά 21 κράτη-μέλη ε, έχουν νομικούς περιορισμούς ε, για το εκλέγει και το εκλέγεστε. Η δημοκρατία που αποτελεί βασικό στατικό του δημοκρατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα είμαι σύντομο, Η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα προτείνει πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα σε βασικού τομεί και κάνουν λόγο και πάλι για τα εμπόδια στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένω. Από την πλευρά έχουμε την ε, νομοθεσία η οποία μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα και στη συνέχεια θα μπορούμε να περιμένουμε τις νέες διατάξεις τις οποίες ε, προετοιμάζει η Επιτροπή για να δουν κατά πόσο μπορούν να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, το να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία ε, και πώς θα συμμετέχουν ε, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ως προς το 2019, η Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων έχει αντιμετωπίσει τα εξή, ότι τα, ε, τα έντυπα με τις πληροφορίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμα ε, για, όλους, ε, τους, για όλα τα άτομα με αναπηρία. Θα επικυρωποιήσουμε το έργο μας σχετικά με την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και προτείνουμε στα τις πολιτικές ομάδες να χρησιμοποιήσετε τις εκθέσεις μας και τα δεδομένα που σας δίνουμε και τις στατιστικές. Έχουμε ε, ενημερωτικά φιλιάδια διαθέσιμα σε όλες τις ε, επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και ε, τον ισότοπο στον οποίο μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο κάθε κράτο Έχουμε Επίσης διάφορα, διάφορες μπροσούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και από τα πολιτικά κόμματα και που ε, δείχνουν πόσο σημαντικό είναι σε πολιτικό επίπεδο να συμμετέχουν και τα άτομα ε, με αναπηρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος. Και τώρα, να δούμε πώς να τον ε, βοηθήσουμε τη λήψη αποφάσεων υπέρ των ανθρώπων με αναπηρία. Μας είπε το Ίδρυμα ε, του Δικαιωμάτων ότι θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα στην άξη του δικαιώματο της ε, ψήφου. Και θα πρέπει να περιορίζεται η δικαιοκρατική ικανότητα για αυτό το σκοπό. Πρόκειται για το άρθρο 12. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει πριν προσχωρήσει κάποιο κράτο σχετική σύμβαση. Δηλαδή η αναπηρία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποστερείται κάποιο από τέτοια δικαιώματα. Πρόκειται για το ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να αναγνωριστεί η ευρωπαϊκή κανένα τους ανθρώπους με αναπηρία. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή στο όσο γίνουν μέχρι σήμερα. Έχουμε διαφορετικά ε, ε, δίκαια και θα πρέπει να δούμε το ότι μέχρι σήμερα υπάρχει μια νομική ρύθμιση, νομικός ε, φραγμός. Θα πρέπει αυτό να έρθει. Θα πρέπει αυτό από την Διεθνή Σύμβαση αυτό να ρυθμιστεί. Άρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αποφάσεις που κατατείνουν σε αυτό που σας προανέφερα. Να δούμε πώς κάπου όπως στην Ανταλουσία θα υπάρχει ένα ίδρυμα με κρατική συμμετοχή οπότε και αυτό το ίδρυμα βοηθά στη λήψη τέτοιων ευμενών αποφάσεων για τους ανθρώπους με αναπηρία. Και έτσι να μπορούν να έχουν αυτονομία α, κίνησης και δραστηριότητας οι άνθρωποι με αναπηρία. με την κυρία Γκράθια Βερνάντεθ Μόγια που συμμετέχει σε αυτό το Ίδρυμα της ε, Φροντίδα των ανθρώπινη εμπειρία στην πόλη της Αλμερίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να σας ε, ενημερώσω για το τι κάνουμε. Πρώτα πρώτα. Για να δούμε. Ποια είναι τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά της επαρχίας μας. Η Αλμερία βρίσκεται στην Ανταλουσία και έχει πληθυσμό 706.690.000 κατοίκων και έχουμε μια ταχεία ανάπτυξη μέσω της γεωργίας. Έχουμε 103 δήμους και υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Έχουμε αρκετούς μετανάστες. Έχουμε μετανάστες από 103 διαφορετικές χώρες. Πρόκειται επομένως για ένα χωνευτήρι διαφορετικών πολιτισμών. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη για οτιδήποτε μελετούμε σε σχέση με την περιοχή μας. Έχουμε στην Ανταλουσία 604.000 που έχουν περισσότερο από 33% αναπηρία. Στην Αλμερία 43.500. Και έχουμε αυτά τα σωματεία που φροντίζουν τα συμφέροντα αυτών των προσώπων μαζί με τις τοπικές αρχές ε, ως επιτοπλής να νομικά πρόσωπα μεικτού χαρακτήρα. Με αυτό το μοντέλο βλέπουμε ότι υπάρχει εγγύηση του πάντα να υπάρχει κάποιο νομικό πρόσωπο το οποίο φροντίζει αυτά τα πρόσωπα ε, που έχουν ε, πολλές φορές περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και που θέλουμε να υπάρχει παντού στην Ανταλουσία. Έχουμε επομένως διάφορες τέτοιες φορείς. Έχουμε μια ομοσπονδία, ε, έχουμε την περιφερειακή οργάνωση, έχουμε και κάποιο φορέα για τα πρόσωπα που έχουν το σύνδρομο Down. Θα πρέπει επομένως να τονίσουμε ότι πρόσφατα έχουμε έναν νέο νόμο. Ή ε, με αυτό τον νόμο αναγνωρίζεται το δικαίωμα του να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικέ υπηρεσίε, τα πρόσωπα με αναπηρία σε αυτό που χρειάζονται. Υπάρχει επίση επίσης ε, νόμος του 2017 ε, που αφορά τα δικαιώματα για τα πρόσωπα με αναπηρία. Έχουμε επίσης προγράμματα, κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλο δράσης, ούτω ώστε να πλησιωθούν αυτά τα πρόσωπα που έχουν αναπηρία ή που α, έχουν εξάρτηση από άλλους για να τα καταφέρουν. Και επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα για πρόσωπα με αναπηρία και πρόγραμμα για γυναίκες που έχουν αναπηρία. Τώρα, η το Ίδρυμά μας συγκροτήθηκε, ιδρύθηκε 4 έκτου του 2007. Δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο σκοπός είναι να προστατευτούν οι ενήλικες που έχουν ε, κάποια ανικανότητα ε, ολική ή μερική από πλευράς νομικής δικαιοπρακτικής ικανότητας και που δεν έχουν συγγενείς να τους ε, πλησιώσουν. Επομένως χρειάζεται υποχρέωση ούτως ώστε κανείς να μπορεί να βοηθήσει την ποιότητα ζωής αυτών των προσώπων για να μπορέσει να τους προστατεύσει τα δικαιώματα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι αριστεία ε, υπάρχει, μπορούμε να υιοθετήσουμε για την διαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και επομένως οι αξίες μας είναι δικαιοσύνη, σεβασμός, ποιότητα, διαφάνεια, ε, όχι στην ε, περιθωριοποίηση και ανεξαρτησία. Είπαμε ότι εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο επιτελεί το Ίδρυμα και πλαισιώνεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς που όμως συνδέονται μεταξύ τους. Κοινωνικό, νομικό και διοικητικό οικονομικό. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα επιτελείο το οποίο είναι πολύ συλλεκτικό και προσπαθούν να προσφέρουν στον καθένα ό,τι χρειάζεται. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι όπως είπατε υπάρχει ένα πρωτόκολλο αναγνωρισμένο. Για κάθε περίπτωση, για κάθε αριστερότητα για όλη την Ανταλουσία. Υπάρχει απόφαση που αναφέρεται στο δικαίωμα του εκλέγην. Και φροντίζουμε το πώς θα βοηθήσουμε κάποιον που έχασε το δικαίωμα στην ψήφο να το ξαναβρει. Αυτά όλα μπορεί να συμβούν στη διάρκεια ζωής κάποιου και άπαξε κάποιο έχει συνέστηση των πρατωμένων, τότε πραγματικά μπορούμε να παραφέρουμε αυτό το δικαίωμα το οποίο χάθηκε. Τώρα, όσον αφορά το πόσους βοηθούμε, και ξεκινήσαμε με 420. Κάθε χρόνο προστίθενται 49 πρόσωπα σε αυτούς που βροντίζουμε και υπάρχουν κάποια νομικά προαπαιτούμενα τα οποία ζητούνται και επεξεργαζόμαστε ε, και νομικά κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το ότι υπάρχει αναπηρία. Έχουμε από όλες τις ηλικίες, ε, προστατευόμενους μεταξύ 40 και 60 ετών και έχουμε και πάρα πολλού αλλοδαπούς από διάφορες χώρες. Όπως είπαμε, σας δώσουμε μια ιδέα για το τι γίνεται σε καθημερινή βάση από το Ίδρυμά μας. Όσον αφορά τα κοινωνικά, ε, μελετούμε κάθε περίπτωση, να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ε, την προσωπικότητα και προσπαθούμε έτσι να έχουμε μεταχείριση σε προσωπική βάση. Να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που καλύπτουν όλα όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο, το οποίο πρέπει να καταλήξει να έχει όσο γίνεται περισσότερη αυτονομία για να μπορεί να ενταχθεί στην ε, κοινωνία. Προσπαθούμε να ε, ενημερώσουμε τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο, να βοηθήσουμε όσον αφορά συντάξεις, παροχές ε, και να βοηθηθεί όσον αφορά κατοικία και απασχόληση και όσον αφορά τώρα τα, ε, τη νομική βοήθεια προσπαθούμε να συντονιστούμε με την εισαγγελία να προστατευτούν αυτό το πρόσωπο από πλευράς ε, νομικής ε, ε κληρονομικά και για την διαχείριση της περιουσίας τους. Τους φροντίζουμε και από πλευράς ε, οικονομικής. Όλα αυτά γίνονται πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων ε, υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά που ακόμα εκκρεμούν και τα έχουν ως στόχους και προκλήσεις πρέπει να προσαρμόσουμε τη νομοθεσία μας ε, στην Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία. Θα πρέπει να αλλάξει και ο, και ο κώδικας για να προσαρμοστεί σε αυτή τη Διεθνή Σύμβαση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα γίνει αυτό. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να γίνει. Να υπάρχει ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων, ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται για τα θέματα των αναπηριών και να υπάρχει ένα ε, παρατηρητήριο ε, για αυτά τα πρόσωπα και για αυτό να λαμβάνουν υπόψη άριστες πρακτικές φροντίδας ε, που να παρέχονται υπηρεσίες συνηγόρου και θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για τις γυναίκες που έχουν κάποια αναπηρία και στρατηγικές. Άρα ακόμα απομένουν πολλά να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Λέω μιλήτρια που τα πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπόρεσε να μεταφραστεί πλήρω. Και τώρα έχουμε τους ε, επόμενους ομιλητές. Hello, my name is Sufyan I'm the e Εγώ Ζακινό και Αλ-Ελαμρανή δηλαδή. Καλησπέρα. μου, Ζακιγιώ. είναι το όνομά μου. Θέλουμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Αναφοράων για την πρόσκληση που μας απίφθηνε. Θέλουμε να μιλήσουμε για τις ε, αναπηρίες και το πώς επηρεάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Χωρίς να επαναλάβουμε ε, όλα αυτά που έχουν ήδη υποθεί, θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, ιδίως όσον αφορά το εκλογικό ε, δικαίωμα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και στην έκθεση της Επιτροπής σας για το CMBRD. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το εκλογικό δίκαιωμα. Τα άτομα με αναπηρίε έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Τα άτομα με αναπηρίε έχουν δικαίωμα να ε, ε, μας πούν τι θέλουν να αλλάξει. Στις εκλογές που έγιναν φέτο, εγώ δεν είχα το δικαίωμα να ψηφίσω, διότι βρισκόμουν υπό νομική κυδαιμονία. Το 2014 όμως συμμετείχα στην εκλογική διαδικασία. Η βελγική διοίκηση ε, της, ε, μου, με ενημέρωσε ότι βρίσκομαι υπονομική κυδαινομία μετά το 2014 διότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ τα, τα χρήματά μου. Επειδή λοιπόν έχω αυτή τη δυσκολία διαχείρισης ε, των χρημάτων μου, μου υπόθηκε ότι δεν μπορώ να ψηφίσω. Μα δεν είναι λάθος αυτό. Ναι, ακούγοντας λοιπόν την εμπειρία του Σοφιάν, θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Άρη Ράς ο υποστηρικτής της Inclusion Europe στις ε, τελευταίες, ε, ε, στην τελευταία εκδήλωση που διοργάνωσε το Ευρωκοινοβούλιο. Τι θα γινόταν αν όλοι έπρεπε να περάσετε ένα τεστ για να έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε. Αν κάποιοι από εσά δεν είχατε το δικαίωμα να έρθετε να προσέλθετε σε αυτή τη σημερινή μας συζήτηση γιατί δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας. Είστε βέβαιοι όλοι ότι θα το παίρνουμε σε αυτό το τεστ. Εγώ αμφιβάλλω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προβληματική αυτή η προσέγγιση. Το να, το να θέτουμε στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και να την αποκλείουμε από την εκλογική διαδικασία. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό. Και ο Επίτροπος ε, Ερμόδιος για ε, Ανθρώπινα Δικαιώματα μας ε, ε, ανέφερε σε σχέση με αυτή την υπόθεση ότι πραγματικά πρόκειται για ε, ε, σοβαρότατη περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο αυτά τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά πολλές φορές δεν απαντώνται με ορθολογικό τρόπο, αλλά με θυμικό. Πολλές φορές, για παράδειγμα, στην, στη Ρουμανία κάποιος θέλει να, να παντρευτεί πρέπει να ζητήσει από τον δικαστή για να βεβαιώσει ότι ε, έχει την δυνατότητα να ε, παντρευτεί. Και τη ρώτησε ο δικαστής τι είναι η αγάπη για σας. Πολλές φορές τα τεστ ε, αφορούν τις γνώσεις γύρω από πολιτικά κόμματα, το, τον κίνδυνο να επηρεαστεί κανείς πολιτικά. Αυτά ήταν τα δύο ερωτήματα. Ποιο εδώ σε αυτή την αίθουσα γνωρίζει τα πάντα για όλα τα πολιτικά κόμματα και ποιο μπορεί να βεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να ε, επηρεαστεί ποτέ από κανέναν. Ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιε εκλογέ αυτό ακριβώ είναι. Μια πυθό μεταξύ ανθρώπων ε, και μια διαπάλη, αν θέλετε, μεταξύ διαφόρων πολιτικών ιδεών. Δεν έχουμε ε, εκτίμηση για το πόσα είναι τα άτομα στην, στην Ευρώπη που στερούνται του εκλογικού δικαιώματο στη βάση τέτοιων διαδικασιών. Στη Γερμανία 80.000 άνθρωποι στερήθηκαν το δικαίωμά τους ε, στις τελευταίες εκλογές. Και ακόμη και η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία μεταξύ του 2013 και 2016 αυξήθηκαν κατά 20.000 τα άτομα που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. 20.000. Από 80.000 στις 100.000 πήγαν οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να το πω αυτό και να επισημάνω και το γεγονός ότι αν σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε το εκλογικό δικαίωμα, να μην ξεχνάμε και μια άλλη πολύ σημαντική διάσταση, που είναι το δικαίωμα του, εκλέγεις, του Βεβαίως, πολύ, με πολύ χαρά ακούσαμε ότι στη Γαλλία οι 50.000 που βρίσκονταν υποκοιδαιμονία πλέον θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαδικασίες. Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν νομικές πράξεις ε, που αποκλείουν τα άτομα αυτά από τον εκλογικό κώδικα τώρα, για στον εκλογικό κώδικα αναφέρομαι, που στερούν από τα άτομα αυτά το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Επίσης, τα άτομα αυτά ε, στερούνται του δικαιώματος της σύστασης ε, νομικού προσώπου, νομικής οργάνωσης. Δεν έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης, δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση, γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Σκεφτείτε το. Οι άνθρωποι με ψυχοκοινωνικές ε, αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν μπορούν να συμμετάσχουν ούτε ατομικά ούτε συλλογικά στην πολιτική ζωή της χώρας τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει πραγματικά να αναδειχθεί. Όπως έχει πει και ο Οργανισμός ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, ο εκπρόσωπος του οργανισμού μάλλον, οι, ε, τα άτομα με αναπηρίες εκφράζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική και για τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα μάλιστα όπου άτομα με αναπηρίες με επιτυχία κατάφεραν να συμμετάσχουν, να στην πολιτική ζωή. Ο Ρόμπερτ Μάρτιν για παράδειγμα απέδειξε μέλος της Επιτροπής CPRD απέδειξε ότι είναι ε, δυνατόν να ε, ε, κατεβαίνει κανείς στην πολιτική και να καταλαμβάνει ακόμα και δημοσιαξιώματα. Πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες συμμετέχουν στη διακυβέρνηση των, των οργανώσεών μας Πολλοί μάλιστα συμμετέχουν και στα διοικητικά συμβούλια. Θέλουμε τώρα να, να επικεντρωθούμε και στην προσβασιμότητα των εκλογικών διαδικασιών. Αυτό τώρα για την προσβασιμότητα στην ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν τα πρόσωπα να γνωρίζουν τι, τι, τι διακύβεται τις εκλογές. Φαντάζομαι αυτό το καταλάβατε λόγω της μετάφρασης, αλλά αυτό ε, είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος γιατί η ενημέρωση δεν σημαίνει ότι κάποιοι με αναπηρία δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπορεί όλοι μας να χτυπηθούμε από την έλλειψη ενημέρωσης. με εδώ έχουμε πάνω από 20 γλώσσες που μιλούνται εδώ. Ε, όλοι μπορεί να υποστούν τέτοια ε, διακριτική μεταχείριση δύο σημαντικά μηνύματα. Θέλουμε πρώτον πληροφορίε για το ποιο μπορεί να συμμετέχει στι ε, εκλογέ, ποιο κατεβαίνει στι εκλογέ. Θέλουμε επίση να διοργανώνεται, να διοργανώνονται συναντήσει με πρέπει τα κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογέ να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα του εκλογικού του υλικού. Κόμματα που ζητούν από του ε, πολίτε την ψήφο του, πρέπει να εμπλέκουν όλους τους ε, πολίτες και τα άτομα με αναπηρία. Τα, οι ευρωβουλευτές πρέπει να μας ακούσουν περισσότερο. Μην μας αποκλείετε από συνεδριάσεις σα. Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Ζητήστε τη συμμετοχή μας. Δεν μας, ενδιαφέρει μόνο, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία, όπως και όλοι οι άλλοι πολίτες μας ενδιαφέρουν ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον, κοινωνικά θέματα, οι εκλογικέ διαδικασίες επίσης θα πρέπει να μας εξηγούνται. Θα πρέπει ε, τα εκλογικά τμήματα να είναι προσβάσιμα σε όλους. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να μας βοηθούν στην άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος. Να εξασφαλίζουν ε, ότι καθένας που θα προσέρχεται στην εκλογική διαδικασία θα έχει όλες τις πληροφορίες. Το 2014 κάτι μου συνέβη. Πήγα να ψηφίσω. Εδώ στις εκλογές που έγιναν στις Βρυξέλλες. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό τμήμα, τους έδωσα την ταυτότητά μου, μου δόθηκε μια κάρτα. Και δεν μου είπε κανείς τι πρέπει να κάνω με αυτή την κάρτα. Οι πληροφορίε για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία δεν ήταν ούτε σαφείς, το παραβάν δεν ήταν ε, προσβάσιμο, έπρεπε να, να κατέβω από το αναπηρικό μου αμαξίδιο και κανένας δεν με βοήθησε, ούτε μου εξήγησε τι πρέπει να κάνω. Ακούγοντα λοιπόν αυτά που λέει ο Σοφιάν, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις ε, θεμελιώδεις συζητήσεις για το πώς θα διοργανωθούν οι εκλογές μέχρι και τις διαβουλεύσεις με τα εθνικά εκλογικά γραφεία πρέπει να εκπαιδευτούν δημόσιοι υπάλληλοι ώστε να βοηθούν άτομα με αναπηρίες για το πώς μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί πολλά από τα μέλη των οργανώσεών μας ε, αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν πώς, πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Πολλά μέλη των αστυνομικών δυνάμεων επίση δεν έχουν λάβει συγκεκριμένη κατάρτιση για το πώ μπορούν να βοηθούν άτομα με αναπηρίε και σε εκλογικέ διαδικασίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην εφαρμογή της CPRD μέσω ε, της ε, διευκόλυνσης των ατόμων με αναπήρες στην ε, συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες. Οι εκλογές λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε στα άτομα με αναπηρία ότι στην μελλοντική Ευρώπη έτσι όπως θέλουμε να διαμορφωθεί όλες οι γνώμεις όλων των πολιτών έχουν αξία. Λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, ε, πέντε λεπτά για ερωταπαντήσεις. Okay, Mrs. Ward. Κύριε Ward, θα πάρω το λόγο. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές που ήρθαν. Δεν είμαι σίγουρη να έχω κάποια ερώτηση, απλά θέλω να από την εμπειρία μου, γιατί υπάρχουν πολλές καταστάσεις όπου δημοκρατία λειτουργεί. Αλλά κάποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία. Προτού, λοιπόν, γίνω πολιτικός και έρθω εδώ, εργαζόμουν σε μια μικρή κοινότητα στην Βόρεια Αγγλία, που αποφάσισε να κάνει ένα συμμετοχικό προϋπολογισμό, κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον σαν ε, project, γιατί αποφάσιζε ο κόσμος πώς θα κατανεμηθεί ο προπολογισμό ε, της κοινότητας. Οργανώθηκε λοιπόν αυτή η ενέργεια. Η ψηφοφορία λοιπόν έγινε μια μέρα που χιόνιζε τόσο πολύ ώστε δεν ήταν προσβάσιμο το μέρος. Επίσης οι ε, συγκοινωνίες είχαν να μειωθεί, είχαν αραιώσει εξαιτίας περικοπών. Έτσι, πολλοί δεν είχαν πρόσβαση στην συμμετοχική, σε μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα Εκτιμώ πάρα πολύ όλα αυτά που είπατε, γιατί θεωρώ ότι αν το καταφέρουμε αυτό σε οποιοδήποτε επίπεδο θα πρέπει αυτή την πληροφορία να την ε, μοιραστούμε και με τα υπόλοιπα επίπεδα της των δημοκρατικών διαδικασιών. Για να κληρώσω λοιπόν ω προς αυτό που έγινε, ήξερα ότι πολλά άτομα με ανεπηρία δεν μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και υπήρχαν ε, άλλα προγράμματα στο σύστημα, οι οποίοι δεν μπορούσαν ε, πάλι να συμμετέχουν. Έχω δει την οργή πολλών ατόμων στο facebook. Έτσι λοιπόν, επικοινωνήσα και της πω ότι μπορείτε να ε, παραπονεθείτε, αλλά ήταν ήδη τόσο κουρασμένοι και εξαντλημένοι από το να πολεμάνε το σύστημα που ήταν τόσο άδικο, ώστε δεν είχαν διάθεση να α, καταγγείλουν τα γεγονότα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ. Γιατί έλαβα δράση για αυτό που είχε γίνει τότε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει σε διάφορες καταστάσεις ε, και, σε, και με πολλούς τρόπους επίσης. Είδα πολλά από το ενημερωτικό υλικό που ε, παρήγαγε το ε, Inclusion Europe για τις ε, εκλογές, το εκπαιδευτικό υλικό για την πολιτική εκπαίδευση, για τους πολίτες, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, χρήσιμα για τους πάντες, γιατί πολλοί δεν έχουν ιδέα, κανείς δεν, δεν, δεν λαμβάνει εκπαίδευση στην πολιτική αγωγή. Γι' αυτό συνέβη και το Brexit. Πολλέ από τι ομάδε ε, ε, με άτομα με, ε, αναπηρία, έχουν περισσότερε γνώσει. Ξέρω περισσότερα από άτομα που για δεκαετίε δεν είχαν εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι προ όφελο όλων μα και ότι μπορείτε να διδάξετε πολλά πράγματα και σε άλλα άτομα για το πώ μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ καλό το πληροφοριακό σας υλικό και θεωρώ ότι είναι... Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας και την ευκαιρία που μου δώσετε να πω την προσωπική μου εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια απάντηση, ενδεχομένως μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ξεφύγει χρονικά. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Δημητρακόπουλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίσετε το ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία που δεν έχουν την νομική ικανότητα, δεν έχουν νομική ικανότητα γενικότερα. Πέρα από τις συγκεκριμένες μορφές νομικής ικανότητας στις οποίες αναφερθήκαμε. Ευχαριστώ. Αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμες γιατί τα κράτη-μέλη δεν συλλέγουν τα δεδομένα και αξιόπιστα δεδομένα για τόμα που στερούνται των ε, δικαιωμάτων τους εξαιτίας της νομοθεσίας. Έχουμε συμπεριλάβει κάποιες ε, αναφορές στην έκθεση του 2014 και στην επικαιροποίηση αυτής της έκθεσης θα κάνουμε κάποιες προβλέψεις όταν θα κάνουμε αξιολόγηση για την κατάσταση χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 34.000 ε, και άτομα στη μία χώρα και τόσα άτομα στην άλλη χώρα. Ένα βασικό συμπέρασμα για να γνωρίζουμε τα άτομα που θα στερούν το δικαιωμάτων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο πάνελ θα το μοιραστούμε. Θα το διευθύνει η Ρώσα Εσταράς. Το θέμα είναι οι γυναίκες με αναπηρία. Buenas tardes, empezamos. Καλησπέρα, σας αυτό το δεύτερο πάνελ, το οποίο είναι αφιερωμένο στις ε, γυναίκες με αναπηρία. Θα πρέπει να αναφέρω όμω ότι στην Επιτροπή για τις υποθέσεις γυναικών ε, τώρα επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο, ένα ψήφισμα που είμαι η συγγήτρια. Αφορά ακριβώ αυτό το θέμα. Και έχουμε και κάποια προφορική ερώτηση. Αύριο θα ψηφίσουμε για αυτό το μεγάλο κείμενο. Ελπίζω πριν γίνει ψηφοφορία να το βελτιώσουμε. Και αυτό θα γίνει σήμερα. Πάντως, τέλος Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου θα υποβληθεί στην Ολομέλη αυτό το κείμενο. Όσον αφορά τώρα αυτές τις γυναίκες, το θέμα έρχεται σε ζωστή στιγμή, γιατί και στην Επιτροπή των Αφορών έχουμε πολλές αναφορές για τα προβλήματα που συζητήθηκαν στο προηγούμενο πάνελ για την προσβασιμότητα, για τα πολιτικά δικαιώματα αυτών των γυναικών. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις διπλή δυσμενή διάκριση που υφίστανται αυτές οι γυναίκες. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το ότι είναι αόρατες. Δεν υπάρχουν κάποιες ε, κάποιοι φορείς και οργανώσεις. Στην Ισπανία έχουμε την Θέρμη. Θα μας τα εξηγήσετε η κυρία τώρα που είναι στο πάνελ. Φραγμή γνωστή σε παιδεία, εργασία, στα ψηφιακά, στις μεταφορές, αλλά υπάρχουν και φραγμοί αόρατοι. Είναι τα εμπόδια εκείνα τα οποία γίνονται αιτία να είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην φαίνονται από κανέναν αυτές οι γυναίκες. Οπότε, η ευρωπαϊκή στατική για αυτές τις γυναίκες ή τέλο πάντων θα πρέπει επιτέλους και η πολιτική ανισότητα ανδρών και γυναικών να καλύψει και αυτές τις γυναίκες λείπουν τα στατιστικά, λείπουν τα δεδομένα. Έτσι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Έχουν πολλοί αξιόλογες εισηγήτριες. Αυτά θα συζητήσουμε. Υπάρχουν κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα, υπάρχει απομόνωση πολύ συχνά, ε, υπάρχει απασχόληση ευάλωτη, περισσότερο από τις γυναίκες παρά από τους άνδρες. Οπότε καταλήγουν σε μία αξιοπρεπή σύνταξη. Και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες γυναίκες που πέφτουν στη φτώχεια όταν ε, μεγαλώσουν. Έχουμε επίση ε, στήρωση αναγκαστική, ε, υποχρεωτική άμβλωση, γενικά υπάρχει δυσμενή διάκριση ακόμα και ενώπιον του νόμου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για τις πνευματικές διανοητικές ασθένειες. Αυτό ε, στο παρελθόν ήταν ένα στίγμα. Αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει περιθωριοποίηση και στην παιδεία. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να τα σκέφτονται όλα αυτά. Θα πρέπει να προβλέπουν ε, την πρικοδοσία για όλα αυτά. Όλα αυτά θα κάνουν πολύ ενδιαφέροντα τα σώδα ακούσουμε από τις προσκεκλημένες μας. Μου λένε, όσον αφορά η δραστηριότητα είναι για αυτή την υπόθεση, ότι στην Περιφερειακή Επιτροπή στους κανονισμούς για κατανομή των ε, πόρων από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία. Οι κανονισμοί αυτοί λέω ότι θεωρείται ως προϋπόθεση για να υπάρξει χορηγία ε, το πρόγραμμα ή το έργο να είναι προσβάσιμο. Θα πρέπει αυτό να τηρηθεί, να μην καταργηθεί, ως προϋποδοσία θα είναι βήμα προς τα πίσω. Έχουμε εδώ και τον φορέα για τους τύφλους. Τον ΟΝΦΕ. Να δούμε τώρα την πρώτη μας προσκεκλημένη. Είναι η ε, Αμάλια. Η Αμάλια Διέγκης. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας αλλά επίσης έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό τον φορέα για την εκμάθηση από απόσταση. Και ασχολείται επίσης με διανοητικές παθήσεις και ασχολείται και με τον φορέα αυτόν που είπαμε, το Ίδρυμα Θέρμη για τις γυναίκες. Ξέρω αυτόν τον φορέα. καλύπτει επιμέρους άλλους φορείς που ασχολούνται με τα πρόσωπα που έχουν αναπηρία. Η πρώτη οργάνωση στην Ισπανία. Αμάλια, ευθύσαμε όσο έχεις τον λόγο για να μας κάνεις την εισηγησή σου. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για τη συνέδεφο που ανέφερες, δεν μπόρεσε να έρθει. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια που εκπρόσωπουμε. Σε όλη την Ευρώπη υφίστανται όλες αυτές τις ζημινές διακρίσεις που μας είπες λόγω φίλου και λόγω αναπηρίας. Είναι ένας οργανισμός Θέλουμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε οι γυναίκες μεγάλες και μικρές να έχουν τις συνθήκες που πρέπει να μπορούν να απολάβουν των δικαιωμάτων τους όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως αναφέραμε απόψε υπάρχει και η Διεθνής Σύμβαση που φροντίζει για αυτόν τον σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει αυτή την Διεθνή Σύμβαση και το άρθρο 6 αναφέρεται στις γυναίκες με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρήσει ότι είναι οριζόντιος αυτός ο στόχος για όλες τις πολιτικές επομένως. Να λάβει υπόψη και τη διάσταση του φύλου όσον αφορά τις ε, ανισότητες. Και έτσι να προωθηθούν τα δικαιώματα αυτών των γυναικών. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί παρακολούθησης της σημειούμενης πρόοδου. Και αυτά να καλυφθούν και από το συνεργατικό κίνημα αυτών των γυναικών. Έχουμε οκτώ χώρες που έχουν τέτοιες οργανώσεις. και έτσι μπορεί να βρεθούν συνομιλητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται είναι να προωθηθεί η έρευνα, κάποιο είδους αρχείο μητρό πληροφοριών, κάποιοι δείκτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το τι γίνεται με αυτά τα πρόσωπα, τι γίνεται με α, τους φορείς τους και να υπάρχει ε, κατηγοριοποίηση ε, όσον αφορά το που ζουν, την ηλικία τους, το φίλο τους. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει επί τη βάση των προβλέπει αυτή η διεθνής σύμβαση, στρατηγικές και οδηγίες να υπάρξουν. Για την ισότητα ευκαιριών, απασχόληση, παιδεία, ίσες ευκαιρίες και για τις γυναίκες με αναπηρία. Αυτή η άποψη, αυτή η οπτική γωνία είναι θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσμενείς διακρίσεις. Είναι και το άρθρο 36 επίσης της Σύμβασης για τα θέματα της δικαιοσύνης. Χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές θα πρέπει να περάσουν τα κατάλληλα μέτρα να λυθούν τα προβλήματα σε όλα τα κρατημέλη να υπάρχει ενημέρωση και όσων δουλεύουν στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί που υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ατιμορρησία πια για ένα σώρο εγκλήματα επί τη βάση του φίλου, Εις βάρος δηλαδή των γυναικών. Οι δεν έχουν προσβασιμότητα, εξαρτώνται από κάποιους που μεσολαβούν. Έτσι δεν προστατεύονται αρκετά τα δικαιώματά τους. Έχουμε επίσης και το άρθρο 17 το οποίο αφορά την προστασία της προσωπικής ακαιρεότητας και αφορά την καταγγελία συμπεριφορών εις βάρος αυτών των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αναγκαστική ε, στηρότητα και ε, όσον αφορά επίσης την αναγκαστική άμβλωση. Ε, επίσης, σε σχέση με αυτό, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει για το άρθρο 23 όσον αφορά την ε, οικογένεια και τον οικοκυριό. Γυναίκες, άνδρες, παιδιά με αναπηρία δεν πλαισιώνονται αρκετά από την πολιτική επασχόληση της Ένωσης. Η νομοθεσία δεν είναι συνεπής. Υπάρχει μια ιεραρχία όσον αφορά τις διαφορετικές μορφές διάκρισης. Και όσοι έχουν αναπηρία προστατεύονται κατά της δυσμενής διάκρισης μόνο στην κατάρτιση και την απασχόληση. Για άλλους λόγους, όπως ας πούμε η φιλή η προέλευση δεν υπάρχει προστασία. Άρα χρειάζεται μια νέα οδηγία που θα διευρύνει την προστασία και σε άλλους τομείς. Στα κοινωνικά επιδόματα, την υγεία και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών του 2010 δεν καλύπτει αρκετά τα δικαιώματα γυναικών και άρα θα πρέπει να υπάρξει καινούρια κατεύθυνση, καινούρια ρότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συγκεκριμένα προβλήματα αυτών των προσώπων, να υπάρξει πιο ενεργή πολιτική και να προωθηθεί πραγματικά η ισότητα των φύλων. Όσον αφορά την βία των γυναικών, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην ε, συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης της Κωνσταντινούπολης. Και Χρειάζεται χρηματοδότηση για να επεξεργαστούμε και να ερευνήσουμε τους δείκτες του τι γίνεται για άνδρες, γυναίκες και παιδιά με αναπηρία σε σχέση με την εκδήλωση βίας εις βάρος τους. Έχουμε ένα σωρό ανθρωποκτονίες σαν συνέπεια της βίας κατά των γυναικών. Να δούμε και το θέμα της κακομεταχείρισης. Επίσης το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει κατάρτιση για την ε, πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά γυναικών και ανδρών αναπήρων. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μελέτες, να φωτιστεί το τι ισχύει, ποια είναι η πραγματικότητα για την στήρωση των ε, αναπήρων σε πολλά κρατημέλη, τι γίνεται με την αναγκαστική και θεραπευτική στήρωση. Δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει αυτή την προοπτική, αυτή την οπτική γωνία της αναπηρίας στην πολιτική υγείας. Και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν μπορεί να ασκηθούν από πολλές από αυτές τις γυναίκες. Επομένως, βλέπουμε ότι τους στερείται και η επιλογή της μητρότητας. Αυτές οι γυναίκες υφίστανται όπως είπαμε στήρωση και αυτό αφορά την ελευθερία επιλογής τους και τον ελεύθερο καθορισμό του τι θα κάνουν για την ε, σεξουαλική του ζωή. Αυτό αφορά και τους ΛΟΑΔ που έχουν αναπηρία. Αυτό αφορά μετανάστες και εκεί επίσης υπάρχουν δεσμένες διακρίσεις και παρενόχληση. Θα πρέπει να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται όσον αφορά τους αναπήρους, τι γίνεται με την ανισότητα και στον τομέα της υγείας, που είναι πολύ χτυπητές αυτές οι ανισότητες, λόγω φύλου. Να προσεχθούν επίσης και αυτοί που έχουν δυσκολία επικοινωνίας, πρόληψη και πλαισίωση υγειονομική σε πλαίσιο προσβάσιμο και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έχουν ε, αναπηρία και σε όσους έχουν δεσμενή θέση λόγω του φίλου τους. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε με το δεύτερο πάνελ. Να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Και εγώ να καταλάβω καλύτερα κάποια πράγματα για, σε σχέση με το ψήφισμα που έχουμε όπως σας είπα. Και τώρα, η κυρία Παπα-Νικολάου. Πελαγία Πούλα Παπα-Νικολάου, που είναι διδάκτωρο εγκληματολογίας στο Εθνικό Καπιτοστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το και ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία. Όλα αυτά θα μας τα εξηγεί στα πλαίσια αυτού του πάνελ όσον αφορά τη δουλειά του πάνελ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ, μεταξύ σας, ανάμεσά σας. Ε, εγώ θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα των γυναικών με αναπηρίες και σκοπός της παρουσίας μου είναι να δώσω έμφαση σε δύο θεματικούς τομείς που είναι η πρόσβαση των γυναικών με αναπηρίες σε ιατρικές υπηρεσίες, στην ιατρική περίθεληση και το άλλο είναι η θυματοποίηση των γυναικών με αναπηρίες, δηλαδή οι γυναίκες με αναπηρίες ως θύματα. Και αφού σας παρουσιάσω τη βάση, θα προχωρήσω σε μια σύνοψη και σε κάποιες συστάσεις πολιτικής για το μέλλον βάση της συζήτησης. Σύμφωνα με την κοινωνιολογική θεωρία για την αναπηρία, οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν διπλό στίγμα. Το να είναι κανείς γυναίκα και ανάπηρη σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί στους ρόλους που έχουν καθοριστεί με βάση πρότυπα άνδρες μη ανάπηρους. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες αποκλείονται από, την, από τις γενικές συστάσεις αλλά και από τις ε, πολιτικές ε, στον τομέα του φεμινισμού, της πολιτικής για τις γυναίκες. Πρώτον, σε σχέση με την πρόσβαση των γυναικών με αναπηρία σε ιατρικές υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι η αναπηρία αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, γενικά αναγνωρίζεται ως ιατρικό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι στην καθημερινότητά μας ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μια γυναίκα με αναπηρία μπορεί να μιλήσει στην καθημερινότητά της, στον οποίο μπορεί να εκφράσει τη σκέψη τη, είναι γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστούν ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία. Πρώτον, χρειάζεται να, να παρέχονται πληροφορίες σε αυτές τις γυναίκες. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να αποφασίσει αυτόνομα για τη δική της ζωή αν θέλει, για παράδειγμα, να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο ή σε έκτρωση. Θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις περιστάσεις, να έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες, ώστε να μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή της. Το άλλο θέμα σχετίζεται με την προσβασιμότητα των κτηρίων, των κτηριακών εγκαταστάσεων των νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας, θα πρέπει τα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις αυτές να μπορούν να είναι προσβάσιμες και από γυναίκες με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ε, σήματα, ε, πινακίδες, ε, ηχητικές πύλες που θα πρέπει να συνοδεύουν όλες τις ιατρικές διαδικασίες και εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι γυναίκες με αναπηρίες όταν επισκέπτονται τέτοιου είδους ιδρύματα, τέτοιου είδους ε, εγκαταστάσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι γενικά προσβάσιμα από όλες τις γυναίκες και από τις γυναίκες με αναπηρίες. Και η τελευταία διάσταση σχετίζεται με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση του ιατρικού ε, προσωπικού, των επαγγελματιών υγείας. Σε αυτή την εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να παρελαμβάνεται ε, και η ενημέρωση των ε, επαγγελματιών της υγείας για τις υποστηρικτικές βοηθητικές τεχνολογίες που βοηθούν πολύ όταν χρησιμοποιούνται σε γυναίκες με αναπηρίες, όταν για παράδειγμα υποβάλλονται σε κάποια εξέταση, σε κάποια ιατρική εξέταση. Ο άλλος θεματικός τομέας αφορά τις γυναίκες ως θύματα. Εγώ, ξέρετε, στη διδακτορική μου διατριβή ασχολήθηκα με τη θυματολογία και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να προτείνω σχετίζεται με τα στατιστικά δεδομένα. που πρέπει να τηρούνται, να συλλέγονται καταρχώς, καταρχάς. Γιατί αυτά μας βοηθούν στον καλύτερο σχεδιασμό της πολιτικής μας, της πολιτικής αντιμετώπισης εγκληματικών πράξεων αλλά και της πρόληψης εγκληματικών πράξεων κατά γυναικών με αναπηρίες. Πολύ λίγα είναι τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και πολλές φορές τα δεδομένα αυτά αφορούν ε, συγκεκριμένες ομάδες γυναικών με αναπηρία. Κοφές, τυφλές, αλλά δεν έχουμε γενική εικόνα. Το δεύτερο σχετίζεται με την ανάγκη ποινικοποίηση ορισμένων μορφών βίας κατά γυναικών. και ορισμένων εγκληματικών πράξεων εναντίον γυναικών με αναπηρία. Όπως είναι για παράδειγμα η στήρωση, η διενέργεια ιατρικών πειραμάτων, η βία ε, υπό ιδρυματικές συνθήκες. Η άλλη διάσταση που θέλω να δείξω είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2012 κάθετος 29 που είναι μια οδηγία στην οποία συμπεριλαμβάνονται διατάξεις με στόχο την παροχή στήριξης σε θύματα βίων εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν κατοχυρώνεται το δικαίωμα των γυναικών με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στο σύστημα της ε, ε, απονομής δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να παρακολουθήσει πιο στενά την εφαρμογή αυτού του άρθρου ώστε να διαπιστώσουμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Η, προσβασιμότητα λοιπόν στο σύστημα δικαιοσύνης προβλέπει και απαιτεί να υπάρχουν προσβάσιμες διαδικασίες όταν εξετάζονται ως μάρτυρες ή ως θύματα γυναίκες με αναπηρίες και οι διαδικασίες αυτές μπορούν ή πρέπει ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνουν ε, ε, διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, ε, στήριξης από ειδικευμένους ε, επαγγελματίες, ψυχολόγους για παράδειγμα, εν γέννη καταρτισμένους ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τα θύματα αυτά, ώστε καταρχάς να καταγγείλουν τη βία που έχουν υποστεί και στη συνέχεια να συμμετέχουν στην, ε, στην προβλεπόμενη για όλους τους πολίτες διαδικασία. Η τελευταία διάσταση αφορά με την ανάγκη ε, να είναι προσβάσιμα τα κτίρια στα οποία φιλοξενούνται γυναίκες θύματα βίας. Όλα αυτά συνδέονται με, την, ε, με τη διάσταση της θυματοποίησης των γυναικών με αναπηρίες. Να σας παρουσιάσω και κάποιες γενικές προσεγγίσεις στις οποίες έχω καταλήξει εγώ. Πρώτον, χρειάζεται να υιοθετηθεί μια ευρύτερη αντίληψη για την ταυτότητα φύλου που θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνει και τις λεσβίες ή τις, τις διεμφυλικές γυναίκες με αναπηρία. Επίσης, Τα πολιτικά θέματα που σχετίζονται με τις γυναίκες με αναπηρίες συνδέονται, ε, πρέπει να ενταχθούν στις, στις, στις γενικές πολιτικές συζητήσεις και πρέπει τέλος να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των διανοητικών ε, αναπήρων θα πρέπει να ε, περιλαμβάνονται στους ορισμούς κάθε κειμένου, κάθε νομικού εγγράφου που αναφέρεται στις γυναίκες με αναπηρίες. Πριν τελειώσω, θέλω να σας δείξω τρεις φωτογραφίες γυναικών με αναπηρίες, τις οποίες θαυμάζω. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τις κοιτάξετε και να τις σκεφτείτε. Η πρώτη φωτογραφία δείχνει την κυρία Σάλιβαν και την κυρία Χέλεν Κέλλερ. Η κυρία Σάλιβαν ήταν δασκάλα της ε, κυρίας Χέλεν Κέλλερ Και νομίζω ότι εδώ θέλω να αναφερθώ στο δικαίωμα της, ε, της εκπαίδευσης, στο δικαίωμα της μόρφωσης. Η άλλη φωτογραφία ε, δείχνει την κυρία Άλισον Λάπερ, που είναι Βρετανίδα καλλιτέχνης, ηθοποιός, που υπερασπίστηκε το δικαίωμά της στη μητρότητα. Η μητρότητα λοιπόν και το δικαίωμα στην μητρότητα είναι κάτι που θέλω να κρατήσετε. Και η τελευταία φωτογραφία είναι μια από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες του φωτογράφου Σεμπαστιάν Σολάδο που είναι διάσημος φωτογράφος με πολύ έντονες οικολογικές ευαισθησίες. Εδώ ε, βλέπετε μια ε, γυναίκα από την Πενίν, αν θυμάμαι καλά, από την Αφρική. Και την ε, διάλεξα αυτή τη φωτογραφία, διότι η ζωή συνδέεται ακριβώς με αυτό το δικαίωμα στη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή σας Σας ευχαριστούμε Πελαγία. Έχουμε άλλα πέντε λεπτάκια, εφτά. Μετά θα τελειώσει η διερμηνία γιατί στις 6.30 τελειώνει το ωράριό τους. Υπάρχει μήπως κάποιος που θα ήθελε να θέσει ένα ερώτημα, κάποια, κάποια παρατήρηση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πραγματικά και εγώ είμαι υπέρ της ε, μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή. Μιλάμε και για το θέμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Πρόσφατα στο αεροδρόμιο σε κάποια πτήση μάλλον ε, συνάντησα τη διευθύντρια της ε, ε της παιδιατρικής κλινικής των Βαλεαρίδων. Εγώ, ξέρετε, ε, είμαι χείρα. Εάν μείνει έγκυος η κόρη μου, δεν τα καταφέρω. Δεν μπορώ να τα ακόμα ένα στόμα. Δεν μπορώ. Ε, έχω κάποιο σύντροφο και επομένως δεν μπορώ, δεν μπορώ να προσθέσω άλλο μέλος στην οικογένεια. 50% επομένως γενετικά υπάρχει η πιθανότητα να επαναληφθεί αυτή στην επόμενη γενιά αυτή η αναπηρία. Οπότε έτσι πάμε στο θέμα της αναγκαστικής στήρωσης. Τι να πω εγώ σε μια μάνα που μου λέει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά μέτρα εναλλακτικά. Τι θα κάνει κανείς άμα είχε τέτοιο παιδί με αναπηρία. Θα πήγαινε εκεί ή θα έκανε κάτι άλλο. Όχι, δεν πρέπει με τίποτα η αναπηρία να οδηγεί σε δυσμενή διάκριση. Ε, όλα αυτά τα οποία είπε αφορούν την ίδια, δεν αφορούν την κόρη της, η κυρία αυτή. Φεραγκούτ. Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την πείσω, γιατί μου έλεγε για μια ζωή καινούργια. Α, εδώ είναι. Η κυρία Στίβενς. Αλλά χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα, φορτισμένα συναισθηματικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη σε επίπεδο συναισθηματικό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν ξέρω, η Χέλγα ε, θέλει να μας πει δύο λόγια. Και μετά η Πελαγία. Πελαγία, πες μας εσύ. Έχουμε τέσσερα λεπτάκια. Πελαγία πρώτη. Το μόνο πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι δεν χρειάζεται μόνο πληροφόρηση για τις συνέπειες της έκτρωσης ή της στήρωσης, αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Π.χ. μια γυναίκα που θα δώσει ζωή. Θα πρέπει να τα γνωρίζει αυτά, γιατί πολλές φορές οι γιατροί δεν ενημερώνουν επαρκώς τους μελλοντικούς γονείς ως προς την αναπηρία, τη λειτουργικότητα και τις ρεαλιστικές διαστάσεις της κατάστασης. Γι' αυτό πολλές φορές οργανισμοί, οι επιτροπές δεν μπορούν να ε, πούν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Άρα το καλύτερο εργαλείο είναι η ενημέρωση για το παιδί που ενδεχομένως θα γεννηθεί ή για την γυναίκα και όλα αυτά είναι φυσικά περίπλοκα ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του σχετικά με αυτό το θέμα για τις γυναίκες με αναπηρία σχετικά με την επιβαλλόμενη στήρωση είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αν το δούμε από διαφορετικέ ε, οπτικέ γωνίε δεν θα έλεγα να πω ότι είναι σωστό ή ότι είναι λάθος, όμως θεωρώ ότι είναι σημαντικό όλοι μας να προσπαθούμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι οι γιατροί αποφασίζουν πράγματα για εμάς και αυτό θεωρώ ότι είναι θεμελιωδώς άδικο. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να συζητηθεί ε, στο πλήσιο της κοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Όχι να συζητάμε τι θα κάνουμε με αυτούς, αλλά να τους συμπεριλάβουμε αυτούς, να τους ε, καλέσουμε στον διάλογο. Άρα το ερώτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξή. Ή σαν με το να αναθρέψεις ένα παιδί. Θεωρείς ότι έχεις αρκετή στήριξη και την απαραίτητη ικανότητα για να αναλάβεις αυτή την ευθύνη. Άρα λοιπόν πρέπει να το συμπεριλάβουμε στη δικασία. Καταλαβαίνω ότι οι γονείς είναι αυτοί, ειδικά όταν κάνουμε λόγο για γυναίκες με διανοητική αναπηρία. Ξέρω κάποιους που είναι παιδιά γονέων με διανοητική αναπηρία και έχουν πει ότι ήταν πολύ δύσκολη η ζωή τους γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς να τους φροντίσουν. Άρα είναι ένα πολύ ευαιστό και πολυπλοκό θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και όχι κάτι που θα εναπόκειται στο, στους γιατρούς ώστε να αποφασίζουν μόνο αυτή την είναι σωστό για τους ασθενείς τους. Θεωρώ ότι το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια με οργανώσεις για τα άτομα με θα πρέπει να ε, κάνουν ακροάσεις, να οργανώσουν συνεδριάσεις. Δεν είναι ένα θέμα απόλυτο. Γιατί με την απόκτηση παιδιών έρχονται και πολλές ευθύνες. Πολλοί ενδεχομένω να μην εκτιμούν αυτόν τον τόνο όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Για μένα όμως το σωστό είναι να το συζητήσουμε με τα άτομα τα οποία θίγονται άμεσα. Τα άτομα με αναπηρία, η θυματοποίηση των ατόμων, των γυναικών με αναπηρία. Το σκεφτόμουν και αυτό το θέμα γιατί όπως πολύ γνωρίζετε. Υπάρχει το Me Movement, το hashtag. Πότε δεν έχετε ακούσει μια γυναίκα με αναπηρία να είναι κομμάτι αυτού του κίνηματος δεν ασχολείται κανείς με τις γυναίκες με αναπηρία. Φυσικά και αυτές έχουν πολύ ψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν, γιατί το δικαστήριο δεν είναι προσβάσιμο για αυτές, ούτε η αστυνομία. Ε, τα μέρες τα οποία μπορούν να βρουν ε, καταφύγιο, ούτε αυτά είναι προσβάσιμα. Γνωρίζω πάρα πολλές ιστορίες παρενόχλησης στο Βέλγιο και σε άλλα μέρη, τα οποία τα σπρώχνουν κάτω από το χαλί ουσιαστικά και τα συγκαλύπτουν. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους και να έχουν την στήριξη που χρειάζονται στη Φλάνδρα. Έχουμε άτομα με τα οποία μπορεί κανείς να επικοινωνήσει, όμως ε, δεν είναι τόσο βέβαιο κατά πόσο αυτό είναι αποτελεσματικό, γιατί υπάρχουν, ε, γιατί οι οργανώσεις θέλουν να κρατήσουν το καλό τους όνομα. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν το διάλογο για να δούμε τι γίνεται ειδικά όταν κάνουμε λόγο για γυναίκες με αναπηρία, γιατί αυτές είναι οι πιο ευάλωτες. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ.